Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Bonjour, chers collègues. Euh, nous, euh, nous allons donc... Euh, Καλημέρα σας λοιπόν. Άρχεται η τρίτη ενότητα συζητήσεων της Μεκτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μας για την 71η, συγγνώμη, 72η σύνοδο. Οι προσκεκλημένοι μας έχουν καταφτάσει σχεδόν όλοι. Βλέπω τον κύριο Ντεμπρόερ που εκπροσωπεί εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Οκτάη κάπου εδώ γύρω θα είναι σίγουρα και δεν θα αργήσει φαντάζομαι. Και πρωί πρωί έχει έρθει ο πρωταγωνιστής ε, καλεσμένος μας, για το πω έτσι, ο κύριος αλχατίπ, ε, πρώην πρόεδρος της Συριακής Συμμαχίας ε, των Αντιφρονούντων και της Επανάστασης μέχρι πολύ πρόσφατα. Μέχρι τις 22 Απριλίου ήταν πρόεδρος. Έχετε προβλήματα διερμηνίας Α, για, για το κανάλι ρωτήστε το Θεό γιατί εγώ δεν ξέρω 26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 Δεν είναι η πρώτη φορά ούτε στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση ούτε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που από την αρχή της σύγκρουσης που είναι πάρα πολλοί μήνες πλέον στη Συρία η κατάσταση στη Συρία και οι ευθύνε και η πολιτική πρωτοβουλία που θέλουμε να ληφθεί και από τις χώρες της περιοχής αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα ε, συζητώνται. Και μεταξύ μας την περασμένη φορά, αν θυμάστε, είχαμε δεχθεί τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον κύριο Νταβουτόγλου, με τον οποίο ανταλλάξαμε απόψεις επί του θέματος. Και πάρα πολύ πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Μαΐου ενέκρινε ψήφισμα, το τρίτο παρακαλώ. Πέντε συζητήσεις έγιναν, τρία ψηφίσματα για το θέμα αυτό. Και πάρα πολύ γρήγορα ζητήσαμε η διεθνή κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινητοποιηθούν όχι μόνο για τα ανθρωπιστικά ζητήματα αλλά και τα ζητήματα προστασίας ε, του αμάχου πληθυσμού. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα ζητήσαμε να ε, ε, εξασφαλιστεί η χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας ε, μιλήσαμε για ανθρωπιστικούς διαδρόμους, ε, για ε, ζώνη απαγόρευσης υπέρπτυσης, για προστασία του πληθυσμού και ζητήσαμε από τα κράτη να αναγνωρίσουν την συμμαχία των αντιφρονούντων ως επίσημο συνομιλητή. Αυτό έγινε. τώρα, μετά από κοινή προσπάθεια Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας, ήρθε μερικός το εμπάργο των όπλων ε, για να ε, επιτρέπεται ε, και η χορήγηση φωνικού υλικού όπως το λένε που ουσιαστικά είναι όπλα. Ξέρω ότι ο προσκεκλισμένος μας ενδιαφέρεται πολύ αυτά τα θέματα γιατί Κατέπληξε το σύμπαν όταν έκανε στι αρχέ του χρόνου πρόταση διαλόγου στον ε, Μπασάρα Λάσαντ. Εμεί υποστηρίζουμε το διάλογο λεγόμενο Γενέβη 2, που από ό,τι φαίνεται η διάσκεψη αυτή δυσκολεύεται να στηθεί. Ε, για να συζητήσουμε για αυτήν την κατάσταση. Ευχαριστούμε τον κύριο ε, ε, Μοαζαλ Χατίμπ που δέχτηκε την πρόταση αυτή. Ε, υπήρξαν δυσκολίες μέχρι τελευταία στιγμή, τις τρεις τελευταίες μέρες ήταν αβέβαιη η έλευσή του. Ε, ίσως ε, πολύ γρήγορα θα δούμε και ένα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ο κύριος Μπέργκερ που πρόκειται να καταφθάσει. Ο κύριος Οκτάη ε, που είναι εκπρόσωπος πολιτικής προστασίας της τουρκικής κυβέρνησης. Καλωσορίσατε αρμόδιος για θέματα επίγουσών καταστάσεων. Και ο κύριος Μπρόουερ είπαμε ότι είναι Διευθυντής Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι μόνο εκπροσωπεί όλος ιδιαίτερο στην ε, Επίτροπό του την κυρία Γεωργίευα που από την αρχή πρωτοστατεί με πολύ στένος ε, και είχαμε την ευκαιρία να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας γι' αυτό. Euh, θα ήθελα τώρα να προτείνω στον κύριο Μόζα Αλχατίβα θέλει να ε, ανοίξει τη συζήτηση, να κάνει την εισαγωγική τοποθέτηση ε, με τα στοιχεία ανάλυσης του, ε, τα αιτήματα που ήταν πάρα πολύ έντονα. Ξέρω ότι έχετε προτείνει και ένα ειρηνευτικό σχέδιο έτσι ώστε να μπορέσουμε στις δικές μας αναλύσεις πλέον και συζητήσεις να συμπεριλάβουμε και τα ανθρωπιστικά θέματα, τα πολιτικά, τα στρατιωτικά και τα θέματα ασφαλείας που πολύ συχνά εμφανίζονται κατακαιρματισμένα στη συζήτηση και ε, ωστόσο συνδέονται πολύ στενά όπως ακούσαμε. Δηλαδή θα πρέπει να ενισχυθεί η στρατιωτική ε, δυνατότητα της αντιπολίτευσης για να μπορέσει καλύτερα από εκεί και πέρα να σταθεί στο ύψος του πολιτικού διαλόγου με τον Μπασάρ Ελλάς. Το ζητήσατε κι εσείς Ήρη και το έχετε θεωρητικοποιήσει μάλιστα. Παρακαλώ κύριε Αλχατίμπ να μας ε, παρουσιάσετε τις απόψεις με πάσα ειλικρίνεια και ελευθερία και χρονική. Όμως μας παρουσιάσετε την κατάσταση παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένως και της ανθρωπιστικής, την οποία δεν ε, υπενθύμησα, τα γνωρίζουμε όλοι, θα μας τα πούν και οι προσκεκλημένοι μας. Ξέρουμε ότι μέρα με τη μέρα είναι όλο και πιο τραγική, πάνω από 4 εκατομμύρια ε, είναι οι εκτοπισθέντες, 1,5 ε, εκατομμύριο οι πρόσφυγες και 100.000 οι νεκροί. Δραματική κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχηθώ καλημέρα σε όλες και όλους και να ε, δηλώσω ότι έχουμε πολύ σημαντικούς προσκεκλημένους σήμερα τον κύριο Ελχατήμ ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Συριακής Αντιπροσωπείας και θα μας ενημερώσει ο κ. Οκτάη που είναι επικεφαλής της ε, πολιτικής προστασίας της Προεδρίας μας ο κ. Ντεμπράουερ της Κομισιόν ο οποίος επίσης θα μας απευθύνει το λόγο σήμερα και θα ήθελα να σας καλωσορίσω, όπως άλλωστε το έπραξε και η συμπροεδρός μου. Στην Συρία σημειώνεται ανθρωπιστική καταστροφή εδώ και καιρό. Έχει έρθει η ώρα να τελειώσει αυτό το ανθρωπιστικό δράμα. Εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Περίπου 100.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία και μόνο έχουμε μισό εκατομμύριο πρόσφυγες σε διάφορα στρατόπεδα ε, προσφύγων τους, ε, στους οποίους έχουμε επιτρέψει να καταλύσουν εκεί 300.000 μόνο στο νότο της χώρας μας προσπαθούν να, προσπαθούμε να βοηθήσουμε η Τουρκία βεβαίως έχει σημαντικό ρόλο να παίξει. Προσπαθούμε πρώτα να υπολογίσουμε πόσο είναι ο αριθμός, πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των ε, σύρων προσφύγων εντός των σύνορων μας. Σίγουρα ο κύριος Οκτάη θα μπορέσει να μας πει λεπτομέρειες εδώ για το πώς θα διαμορφωθεί, πώς διαμορφώνεται και θα διαμορφωθεί η βοήθεια που προσφέρεται στα πρόσωπα αυτά εντός Τουρκίας. Ελπίζουμε ότι το δράμα αυτό στην Συρία θα πάψει κάποια στιγμή. Όλος ο κόσμος, η διεθνής κοινότητα οφείλει να πάρει πιο σοβαρά υπόψη το σοβαρό αυτό πρόβλημα. Εμείς ως συμπρόεδροι θεωρήσαμε σωστό και σημαντικό να εγγραφεί το θέμα στην ημερησία διάταξη έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι χώρες μέλη να επιληφθούν του θέματος, να ακούσουν τις φωνές των σύρων, να ακούσουν τις κραυγές απόγνωσης των παιδιών και να αντιληφθούν ότι φέρουν ευθύνη, την οποία οφείλουν να αναλάβουν. Ελπίζω ότι η σημερινή ε, συνάντηση θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα για την Συρία. Σας απευθύνω λοιπόν το θερμό καλώς ορίσατε σε όλους τους προσκεκλημένους μας, ιδίως τον κύριο Χατίμπ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τη Μεκτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την υπόθεση της Συρίας. Ε, καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι το δράμα αυτό δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία μας. Ε, θα πρέπει να τεθεί ένα τέρμα, αλλιώς θα επεκταθεί. Οι ε, Ηνωμένε Πολιτείε και η Ρωσία, πρέπει να σας πω, ε, ούτε η μία ούτε η άλλη δεν έχουν σαφή ε, εικόνα, σαφές όραμα. Διπλωματικές συζητήσεις γίνονται ιδέες χωρίς πραγματικό όραμα. Οι Ευρώπη μας λέγουν ότι είναι η Ήπειρος που φέρει τη σοφία του κόσμου. Ότι υπάρχει μια σοφία ε, ανάμεσα στις σχέσεις Ευρώπης Μέσης Ανατολής. Πότε αυτή η σοφία λοιπόν θα ε, μεταφερθεί στην πράξη, θα μεταφραστεί ε, σε δράση για να τερματιστεί το δράμα της Συρίας. 50 χρόνια δικτατορία υπέστη η Συρία αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι καινούριο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται στον κόσμο ως ε, νέο, ως πρωτοφανές, αλλά εμείς το ζούμε τα τελευταία 50 χρόνια, σε πιο περιορισμένο ίσως επίπεδο. Ε, ουδέποτε ε, απολαμβάναμε ελευθερία στη Συρία. Ο Συριακός λαός το μόνο που ήλπιζε είναι να μπορεί να κοιμάται χωρίς αυτό το φόβο, χωρίς αυτό το δρόμο. Η δική μας συμμαχία προσπάθησε τα πάντα, όλες τις λύσεις. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος του πολέμου, δεν πιστεύω στον πόλεμο. Πιστεύω ότι ο πολιτικός διάλογος είναι εκείνο που μπορεί να καταλήξει σε αποτελέσματα. Πριν φύγω από τη Συρία, ε, φυλακίστηκα δύο φορές, διότι είχα προτείνει δύο ειρηνικές λύσεις στην κρίση. Το καθεστώς έχει δύο μεγάλα ελαττώματα. Ε, διακατέχεται από ε, μεγάλη υπερηφάνεια και ε, από μεγάλο ψεύδος. Λοιπόν, είναι περήφανοι και ψεύτες και δεν θέλουν και πολιτική λύση. Προσπαθούν πάντα να κερδίσουν χρόνο. Και ποιος τους έχει δώσει αυτή την ευκαιρία και αυτή τη συμβολή μάλιστα. Ακούγεται ότι είναι οι Ρώσοι. Ε, για να καταφέρουν, λέει, ότι κατάφεραν και οι Ρώσοι στον Κρόσνη, στην Τζετζενία. Ακούσαμε για το Στάλιγκραντ ότι έχει ζήσει τρομερή καταστροφή. Ε, εγώ θα σας έλεγα ότι το Στάλιγκραντ οχριά σε σχέση με αυτά που ζει σήμερα η Συρία. Οι επιπτώσεις ε, και οι πληγές από το όσα συμβαίνουν σήμερα είναι τρομακτικές. Σειρά σε λίγο έχει ο Λίβανος. Η Ορδανία ενδεχομένως επίσης. Γνωρίζετε ότι πάνω από 40% των Ιορδανών είχαν πάρει συριακά διαβατήρια. Να σας πω και μια ιστορία. Κάποτε ε, ήταν κάπου ε, κάποιοι μοναχοί χριστιανοί με το Ευαγγέλιο στα χέρια. Ήρθε να τους δύο ηγούμενός τους και τους είδαν να κλαίνε και ε, τους ρώτησε γιατί κλαίτε. Και εκείνοι απάντησαν ε, κλαίμε διότι μας πήραν τα Ευαγγέλια. Και τι ωραία, κάθεστε και κλαίτε επειδή σας πήραν τα Ευαγγέλια από τα χέρια να ψάξετε να τα βρείτε. Τι κάθεστε και κλαίτε. Λοιπόν, ε, σήμερα όλοι καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και κλαίμε. Δεν κάνουμε τίποτα για να ε, σταματήσουμε αυτή την κρίση. Πολιτική ε, λύση επιζητούμε και πολιτική λύση επιδιώκουμε. Και γνωρίζω ότι οι Τούρκοι αδελφοί μας και οι πολίτες της Τουρκίας άνδρες και γυναίκες ενδιαφέρονται για την κατάσταση και ανησυχούν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Δαβούτογλου, επισκεφθεί ήδη έξι φορές στη Συρία. προσπαθεί να βοηθήσει. Έχει πει και στον Μπάσα Λάσαντ τον ίδιο, θα σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε αυτή την κατάσταση, αλλά γνωρίζουμε ότι ε, αψηφείτε τις διεθνείς συμβουλές και τη διεθνή βοήθεια. Ε, το Συριακό καθεστώς βασίζεται σε άγριες πρακτικές σε, ε, στην αμέριστη ε, υποστήριξη του Ιράν και επίσης είναι ένα καθεστώς το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θέλει να χάσει αυτά τα ερίσματα. Ούτε την ηγεμονία και την εξουσία στη χώρα. Ακόμα και οι πιο μετριοπαθείς Αυτά πιστεύουν. Εμείς θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να τους μεταπίσουμε. Ας πούμε, ο στρατηγός Αμπτέλ Φατάχ Κοτσίε που ήταν αρχηγός στρατιωτικής υπηρεσίας ε, ε, ε, πληροφοριών που είναι αλεβίτης και αυτός ήταν και πιο μετριοπαθής από τους υπολείπους. Τώρα είναι υπό κατοίκον περιορισμό ακριβώς επειδή επέδειξε μετριοπάθεια. Οι υπόλοιποι ε, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί είχαν επίσης την ίδια μεταχείριση. Τους καθαίρεσαν όλους για να ε, διατηρηθεί μόνο η σκληρή και άγρια γραμμή δράσης. Αυτά που συμβαίνουν στη Συρία είναι απερίγραπτα. Θα προσπαθήσω να σας δώσω ένα παράδειγμα είχα κρατηθεί σε ένα κελί 15 τετραγωνικά εμβαδών και πάνω από 71 κρατούμενοι, 72 με μένα, στα 15 τετραγωνικά. Και μεταξύ των 72 ήταν ε, κάποιος που είχε παραφρονήσει ε, και, χωρί, και ήμασταν όλοι σε ένα κελί 15 τετραγωνικά 72 άτομα χωρίς ε, κανένα εξαερισμό και κοντέψαμε όλοι να τρελαθούμε γιατί είχαμε ένα παράφρονα μέσα στους 72 σε ένα κελί 15. Είναι το κελί 215, είναι γνωστό, περίφημο. Και υπήρχαν και άλλα κελιά, 10 τετραγωνικά με 30-40 άτομα στιβαγμένα, ε, με ψυχικά προβλήματα. Και κάθε φορά ε, μας έφεραν ένα κρατούμενο ακροτηριασμένο, τον οποίο είχαν τυφλώσει, του είχαν ε, ε, κόψει τα αυτιά και τον είχαν μέσα στα αίματα, ε, μέσα στις ακαθαρσίες και, και σώματα σε σύψη ακόμα, άφηναν ζωντανούς ανθρώπους μαζί με νεκρούς σε σύψη μέχρι και μία εβδομάδα. Και όταν βάζεις κάποιον με ψυχικά προβλήματα σε ένα ε, τέτοιο περιβάλλον με, τόσο κόσμο στιβαγμένο, ε, γίνεται δίμιο των υπολείπων. Και φαντάζεστε, κλείνεται έναν άνθρωπο με τέτοια προβλήματα μια εβδομάδα με τόσο, ε, τόσο κόσμο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θέλω να με ψημυρώ ούτε να κλαφτώ. Είναι βασανιστήρια και αφορούν όλους. Μέχρι και παιδιά βασανίζονται. Και αυτά είναι στίγματα που θα μείνουν στο μέτωπο της ανθρωπότητας, στο πρόσωπο της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει σοβαρότητα στην αντιμετώπιση κατάστασης αυτής από τη διεθνή κοινότητα. Ποιος ήταν ο ρόλος της Ευρώπης για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ ούτε ανεξάρτητη ούτε αυτόνομη στη δράση της. Γίνεται λόγος ε, ε, για ε, εξοπλισμό της αντιπολίτευσης. Η Ρωσία υποστηρίζει το καθεστώς. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ξέρουμε τι θέση έχουν. Και σήμερα γνωρίζουμε ότι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν υπάρχει ομοφωνία για να εξοπλιστεί η αντιπολίτευση. Διερωτώ με, γιατί δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλία ανεξάρτητη για να λυθεί η κρίση. Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν αρκετή ε, ε, εικόνα, δεν έχουν όραμα. Μας προτείνουν τη διάσκεψη της Γενέβης 2, λέει. Για ποιο λόγο και πού θα βασιστεί αυτή, με τι ορίζοντα, με τι όραμα. Γίνεται λόγος για μια συμμαχική κυβέρνηση για να μιλήσει για κυβέρνηση συνασπισμού θα πρέπει να αισθάνεσαι ασφαλής σε μια χώρα για να μπει στην κυβέρνηση. Αυτό δεν συμβαίνει στη Συρία. Το καθεστώς ε, εκτέλεσε το στρατηγό Ραζί Κανάν Υπουργό εσωτερικών. Πώς έγινε αυτό. Ξέρω ότι δεν ήταν κανένας Άγιος καλός άνθρωπος ήταν ε, υπεύθυνο για πολλέ βιαιότητε στο Λίβανο, παρόλα αυτά τον έκαναν Υπουργό Εσωτερικών. Και εγώ λέγω ότι όσο κακός και να ήταν, χρειάζεται έρευνα να διερευνηθεί ο τρόπο με τον οποίο θανατώθηκε. Ο στρατηγός Μοχάμετ Σουλεϊμάν, υπεύθυνο για την ασφάλεια της χώρας ολόκληρη, Επίση δολοφονήθηκε χωρί καμία έρευνα, χωρί καμία ανάκριση, ε, για να βρεθούν οι αιτίε του θανάτου του. Είναι άγριο το καθεστώς εκεί. Η Ευρώπη έχει ιστορικούς δεσμούς, έχει πολύ μεγάλη γνώση και πρέπει αυτόνομα να δράσει, να αυτονομηθεί για να βοηθήσει στην επίλυση αυτής της κρίσης. Προσωπικά ανήθηκα να συμμετάσχω σε πολλές διασκέψεις για πολλούς ε, λόγους. Γίνεται λόγος μόνο για μειονότητες, για τρομοκρατία και για χημικά όπλα. Και τα τρία αυτά ζητήματα χρειάζονται νέο ορισμό. Τρομοκρατία, ακεραιόφρονες ομάδες, φονταμεταλιστές. Στην αρχή της επανάστασής μας δεν υπήρχε ουδής φονταμεταλιστής πουθενά και κανείς εξτρεμισμός στη Συρία. Ο Συριακός λαός αφέθηκε στη μοίρα του όμως ανάμεσα στα χέρια αυτών των δημίων και τώρα ξαφνικά διαρωτώμεθα πώς εμφανίστηκε αυτός ο φονταμεταλισμός. Δεν τους θέλουμε εμείς τους εξτρεμίστες, τους φονταμεταλιστές. Αυτοί καταστρέφουν ε, τις υποδομές και τη δομή της χώρας και του, Ισλάμ ε, εκ των έσω. Ε, δεν τους θέλουμε εμείς αυτούς. Έτσι έχουν τα πράγματα τώρα. Ε, έχουμε ένα λαό που είναι στα χέρια των δημίων του ε, χωρίς κανένα προστάτη. Και υπάρχει και κρατική τρομοκρατία. Ωραία. Μπορεί να υπάρχουν εξτρεμιστικές ομάδες με πρακτικές ε, εξίσου εξτρεμιστικές. Ε, εσείς τι λέτε όμως για αυτό το κράτος, το δρομοκράτη, το οποίο έχει τρομοκρατικές μεθόδους τα τελευταία 50 έτη παρακαλώ. Υπάρχει κάποιος που είναι αλεβίτης, που είναι ε, κοντινός του καθεστώτος και ε, ακτιβιστής και ε, οπαδός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Αλχάι, Αμπτελαζής Αλχάιρ, πήγε στην Κίνα και στη Ρωσία και τον δέχτηκε ο κύριος Λαυρόφ και παρά το γεγονός ότι είναι κοντά, ε, άνθρωπος του καθεστώτος, τον συνέλαβαν γιατί το συνέλαβαν παρόλο που είναι δικός τους, γιατί ε, ε, θέλει να βρεθεί ειρηνική λύση και όχι να είναι χωρισμένη η Συρία με βάση θρησκευτικές κοινότητες. Έχουμε φτάσει σε επίπεδα αγριότητας πρωτοφανή, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια φαινόμενα. θα είναι πολύ ανητική εξέλιξη αν δεν κάνουμε κάτι θετικό. Η πολιτική πίεση, το πολιτικό λόμπι, χρειάζεται να διατηρηθεί. Έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η ε, προμήθεια όπλων από τη Ρωσία. Γιατί αφήνουμε τη Ρωσία να δίνει πυράβλους Patriot, αντιπυραυλικά συστήματα ε, στο Συριακό καθεστώς. Στη Βόρεια Συρία Υπάρχει μια ζώνη που θα μπορούσε να ε, διαφυλαχθεί να γίνει ασφαλής και να ε, βάλουμε εμείς οι στοιχείες Patriot. Οι Τούρκοι φίλοι μας ε, ανέλαβαν μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία και ευθύνη. Αλλά όταν πηγαίνουμε στην Τουρκία δεν θεωρούμε ότι είμαστε σε ξένη χώρα. Μας βοηθούν, μας διευκολύνουν πάρα πολύ. Ξέρω ότι η παρουσία των Σύρων στην Τουρκία δημιουργεί προβλήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας δικά τους. Και σήμερα ε, ε, το καθεστώς ε, της Συρίας εκμεταλλεύεται αυτές τις αντιφάσεις. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ανθρωπιστικός διάδρομος ασφαλής για τη δίωδο των πολιτών, του αμάχου πληθυσμού. Αυτό είναι εύκολο να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε δαπανηρό είναι. Και στο, λέω με κάθε ειλικρίνεια, το επαναλαμβάνω κάθε φορά που έχω την ευκαιρία, το συριακό καθεστώς δεν είναι ένα καθεστώς που διέπεται ας πούμε, από τη θρησκευτική κοινότητα των Λεβιτών και, και κυριαρχούν εκεί. Αυτό είναι πρόφαση. Χρησιμοποιούν ε, αυτή την ομολογία για να στραφούν εναντίον όλων των υπολείπων ε, με σκοπό να παραμείνουν στην εξουσία, με ομότητα, με αγριότητα, με βία. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ ε, λυπημένοι, πάρα πολύ συντετριμένοι για κάθε νεκρό που έχουμε ε, μας γεμίζει θλίψη αυτό. Αλλά εξίσου θλίψη μα γεμίζει όταν σκοτώνεται κάποιο από το άλλο στρατόπεδο. Δεν θέλουμε να κυριαρχεί ο θάνατο. Αυτοί που διοικούν σήμερα τη Συρία, ε, που έχουν βάλει χέρι στη Συρία, είναι ε, εγκληματίε, συμμορία. Τα θύματα μας κάνουμε να ε, θρηνούμε όλα τα θύματα. Το καθεστώς θέλει ε, να γίνει θρησκευτική αυτή η σύγκρουση. Εμείς θα πρέπει να ε, σταθούμε αντιμέτωποι σε αυτό συμπαγής. Δεν, να μην ε, θεωρητικοποιηθεί ο θρησκευτικός χαρακτήρας. Είναι απλώς ένα άγριο καθεστώς ε, ε, στρατιωτικοποιημένο και καθημερινά σκοτώνει τους πολίτες και το λαό. Αν δεν κάνουμε τίποτα τώρα θα ενταθεί αυτό, θα είναι ακόμα μεγαλύτερη έκρηξη και είδαμε τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης και αυτής της κρίσης ήδη να εξαπλώνονται στο Λίβανο. Τα ίδια στην Ιορτανία η Τουρκία ίδια δεν πρόκειται να βγει αλόβητη από την ε, ιστορία αυτή. Και η Ευρώπη με την ιστορία της γνωρίζει ότι η Ρωσία είναι ένα καθεστώς με μια ιδιαίτερη νοοτροπία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θέλουν να εμπλακούν περισσότερο σε τέτοια διεθνή θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ κοντά μας και ιστορικά και γεωγραφικά και μπορεί να δράσει. Πριν από 1,5 μήνα ανελήφθη άλλη πρωτοβουλία. Ο Μπασάρ Λάσατ ε, το είχε περιφρονήσει αυτό το, έτσι, ε, με απαξιωτικό τρόπο ε, το σχολίασε και ξεπερνάει τη διάσκεψη της Γενέβης 2. Στη Γενέβη 2 γίνεται λόγος για κυβέρνηση συμμαχική, έτσι, συνασπισμό του καθεστώτος με την αντιπολίτευση. Ε, δεν γίνεται αυτό. Εγώ μιλώ για άλλη πρωτοβουλία που λέει το εξής. Ο Μπασάρ Ελασάτ να ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί σε δύο ή τρεις μήνες, ας πούμε, αλλά στο μεταξύ θα παραδώσει στο σημερινό Πρωθυπουργό όλες τις εξουσίες. Εμείς δεν θέλουμε οπωσδήποτε να πάρουμε την εξουσία. Αυτό που θέλουμε είναι να φύγει ο Άσαντ. Ας αναθέσει, ε, ας παραδώσει όλη την εξουσία στον Πρωθυπουργό του, τον οποίο ο ίδιος έχει διορίσει. Και ο Πρωθυπουργός να διορίσει από εκεί και πέρα μέτριο παθής για να κυβερνούν τη χώρα. με γενική αμνηστία υπέρ όλων ε, όσοι ε, πολέμησαν στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο. Και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο σημερινός πρόεδρος θα μπορούσε να πάρει και την άδεια να καταλήψει τη χώρα με 500 δικούς του που θα επιλέξει εκείνος. καμία σημασία δεν έδωσε σε αυτή την πρωτοβουλία. Θέλει να γκρεμίσει όλη τη χώρα, να καταστρέψει όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει χωριό που να έχει αφήσει όρθιο αυτό το καθεστώς. Υπάρχει ένα χωριό που καταστράφηκαν 85 φούρνοι. Και κατακρεούργησαν τον άμαχο πληθυσμό γυναικόπαιδα και τα ζήμωσαν μαζί με τη ζήμη στους φούρνους καταλαβαίνετε ότι δεν έχει κανένα φρένο, δεν έχει κανένα ταμπού αυτή η κυβέρνηση, καμιά κόκκινη γραμμή. Μέχρι πότε θα σφάζουν το λαό έτσι. Τσουνάμι θα γίνει αυτή η κρίση και θα καλύψει όλο τον κόσμο. Σας προειδοποιώ. Εκατομμύρια εκτοπισμένους έχουμε εκτός των συνόρων μας αλλά 6 με 7 εκατομμύρια εκτοπισμένους στο εσωτερικό της χώρας. Δεν υπάρχει καταφύγιο. Πολύ εύκολα σκοτώνει κανείς τον κόσμο. Λοιπόν, η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει με συνέργεια, με καινοτομία, με, με, με φαντασία κάπως για να λυθεί αυτή η κρίση. Δεν χρειαζόμαστε διασκέψεις διεθνείς. Οι διεθνείς διασκέψεις τι κάνουν. Ε, ελαφρύνουν τη συνείδηση της κοινή γνώμης, της διεθνούς κοινότητας, ε, αφαιρούν κάποιο βάρος ε, των διεθνών διοικούντων για να μην πάρει κανείς τις ευθύνες του. Ο Συριακός λαός είναι φιλήσυχος λαός, είναι, είναι καλός λαός, ανεκτικός. Θα μπορούσε να είναι ένα θετικό στοιχείο στην ανθρωπότητα αλλά και ένας ε, παράγων ε, που μπορεί να κάνει να κυριαρχεί το χάος παντού. Ευχαριστώ, σταματώ εδώ. Ουφ. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά τα λόγια σας μας τάραξαν. Τα μέλη hm, της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, τι να σας πω, ευχόμαστε όλοι να είχατε ξεφύγει την μοίρα αυτή, αλλά πρέπει όλος ο κόσμος να ακούσει τη φωνή σας, όχι μόνο η Ευρώπη. Αυτή την κραυγή πόνου πρέπει να την ακούσουν όλοι. Το θανατικό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να φύγει ο Ασάντ από την εξουσία. Καταστρέφονται άνθρωποι. Κατά χιλιάδες σκοτώνονται οι άνθρωποι στη Σύρια. Όπως είπατε, Δέκα εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Πεθαίνουν παιδιά, γέροντες, άρρωστοι. Και όμως η ανθρωπότητα τηρεί σιγή. Δεν είναι αποδεκτό αυτό. Στους εκπροσώπους εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχω να πω το εξή. Θα έπρεπε να είναι παρόντε και παρούσε εδώ και να τα ακούσουν τα πράγματα αυτά. Αλλά δεν είναι. Τα μέλη τη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αυτά συζητούνται εδώ, κάτω από την στέγη τη δική σας. Λέτε ότι θέλετε κάτι να κάνετε για αυτή την καταστροφή και δεν είναι κανείς εδώ. Αυτός ο πόνος πρέπει να ακουστεί. Είμαστε στο πλευρό σας. Και ελπίζω, πρώτο Θεός, θα βρούμε λύση. Αλλά η ανθρωπότητα πρέπει να αντιδράσει, να κάνει κάθε τι το δυνατό για να σταματήσει η τραγωδία αυτή. Με κάθε μέσον πρέπει να κινητοποιηθεί. Η κυρία Φλότρα εγκατέλειψε για λίγη ώρα την αίθουσα. Θα δώσω λοιπόν εγώ το λόγο τώρα τον κύριο Μοντισόγλου. Έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακολούθησα προσεκτικά αυτή την ε, ανάπτυξη των πιο πρόσφατων εξελίξεων. Τι αισιόδοξη προοπτική να δώσω τώρα. Είναι γνωστή η δυσκολία της κατάστασης στην ίδια τη Συρία και στην γειτονική περιοχή της. Βρισκόμαστε σε σύγκρουση με πολλούς άλλους παράγοντες και όχι μόνο με τη κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ένα θέμα που είναι ξεκάθαρο είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματική ανθρωπιστική τραγωδία από τις πιο σημαντικές που έχει δει ο κόσμος μέχρι σήμερα. Από την άλλη μεριά η βαρύτητα της καταστάσεως, η βαρύτητα της κρίσης, η ανθρώπινη δυστυχία, οι συνέπειες για τις γειτονικέ χώρες που δεν είναι μόνο οι αριθμοί των προσφύγων αλλά και κοινωνικές συνέπειες που ταράζουν τις λεπτές ήδη ισορροπίες στην περιοχή. Αυτά δείχνουν ότι και βέβαια η ανθρωπιστική υποστήριξη και οι πρωτοβουλίες που ήδη έχει αναλάβει η διεθνής κοινότητα είναι σημαντικές. Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να λύσουμε την κρίση αυτή μοναχά με ανθρωπιστική βοήθεια. Υπήρξατε επικριτικός απέναντι σε ορισμένες πρωτοβουλίες που αναλύθηκαν τους τελευταίους μήνες. Βεβαίως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ από τη μια μεριά των Ρώσων και Αμερικανών. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση παρά μόνο πολιτική και πρέπει πάνω σε αυτήν να δουλέψουμε. Είπατε Μωάς ότι η Ευρώπη δεν έπραξε τίποτε. Εγώ δεν θα ήμουν τόσο επικριτικός. Και δεν θέλω μόνο να αναφέρω την οικονομική στήριξη που ήδη έχει προσφερθεί από τριμήνου. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Ντεμπράουερ, θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες, ίσως να μην είμαστε στο προσκήνιο, αλλά αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και πράττουμε πάντο δυνατό για να φέρουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής λύσης που θα οδηγήσει σε τέλος την βία και θα οδηγήσει σε μια μεταβατική κυβέρνηση. Εκεί βλέπουμε το ρόλο μας εμείς σήμερα. Να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε ώστε να φτάσετε σε αυτή την πολιτική λύση. Ξεκινήσαμε ήδη από την αρχή της εβδομάδος με μια συνολική απάντηση την οποία εμείς αποκαλούμε response to the crisis που έχει διάφορα στοιχεία, διάφορες παραμέτρους με πρωτοβουλίες για να αποφευθεί η κρίση να φτάσει ακόμα περισσότερο στην Ένωση. Και εμείς, όπως είπε και ο Μωάς, βρισκόμαστε σε κρίση. Και η κρίση αυτή είναι σήμερα μπροστά στις πόρτες μας. Για να επιστρέψω σε αυτήν την ε, συνολική απάντηση, αντίδραση είναι μία από τις παραμέτρους της να φτάσουμε σε μία διαρκή πολιτική λύση για την κρίση. Πράγματι, η Γενέβη, η Γενέβη 2, είναι εξαιρετικά δυσχερής διαδικασία και όλοι σήμερα προχωρούν πολύ προσεκτικά. Υπάρχουν βαθιές διαφορές, σημαντικές και βαθιές διαφορές σε ό,τι αφορά ποιος θα συμμετάσχει στη διαδικασία αυτή. Διαφορές σε ό,τι αφορά το ποιος θα πρέπει να προσέλθει και ποιος δεν θα πρέπει να προσέλθει. Διαφορές υπάρχουν ακόμα και μεταξύ της ίδιας της αντιπολιτεύσεως σχετικά με το ποιος θα πρέπει να προσέλθει και ποιος όχι. Από την άλλη μεριά, ρωτώ, έχουμε άλλη λύση, άλλη από το να προσπαθήσουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημιουργήσουμε την πλατφόρμα αυτή η οποία μπορεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο να συμβάλλει στην περάτωση της κρίσης. Αυτό είναι το πλαίσιο λοιπόν μέσα στο οποίο υποστηρίζουμε πλήρως την πρωτοβουλία που ανέλαβαν Αμερικανοί και Ρώσοι. Και πάλι μιλούμε εδώ για εξοπλισμό, για ζώνες απαγόρευσης πτήσεως και μέσα στην Ευρώπη χώρες μέλη τάσσονται υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Είτε μας αρέσει είτε όχι, σήμερα πιστεύουμε ότι η διαρκής ειρήνη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί χωρίς πολιτική λύση στην κρίση. Ποιες είναι οι άλλες επιλογές. η σύγκρουση στην Συρία συνεχίζεται, είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν υπάρχει προοπτική καμιά από τις πλευρές να κερδίσει στη σύγκρουση αυτή και αντιθέτως στην ουσία προκαλεί μια ας πούμε, κληρονομιά εσωτερικών συγκρούσεων που θα συνεχιστούν για πολλά χρόνια. Λίγα λόγια για τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει εδώ και παραπάνω από δύο χρόνια. Πρωτοβουλίες στήριξης του συριακού πληθυσμού, στήριξης των εκτοπισμένων, των προσφύγων, ακόμα και των παιδιών, που σήμερα γιατί μιλούμε για τους πρόσφυγες, μιλούμε για εκτοπισμένους, αλλά δεν μιλούμε για τα μικρά παιδιά που εδώ και τρία χρόνια δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, στη Συρία την ίδια. Και αυτά θα τα δούμε μπροστά μας πολύ σύντομα, τις επιπτώσεις. Πρωτοβουλίες ακόμη για να ενισχύσουμε και τις γειτονικέ χώρες, τις κοινότητες οι οποίες υποδέχονται τους πρόσφυγες στο Λίβανο, στην Ιορδανία, να βοηθήσουμε επίσης να ενισχύσουμε τους θεσμούς εκείνους στο Λίβανο και στην Ιορδανία που πάσχουν τώρα από τους αυξημένους αριθμούς προσφύγων και ένα πράγμα που θα πω ακόμη είναι ότι φτάνουμε σε λίγο στο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στήριξης για την ε, Συριακή κρίση σε ανθρωπιστική και μη ανθρωπιστική βοήθεια. Αν μου επιτρέπετε θα αρκεστώ σε αυτά κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μοντέζογλου να δώσω το λόγο στον κύριο Μπράουερ ε, για να συνεχίσει για την ευρωπαϊκή πολιτική, επειδή βασικά όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, διότι εδώ αντιπροσωπεύεται την Επίτροπο Γεωργίευα, οπότε θα επικεντρώσετε την ομιλία σας ε, σε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις χώρες όπως η Τουρκία που δέχονται τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Προφανώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρέμβει κανείς για αυτό το θέμα αφού άκουσε τον κύριο Αλκατίμπ. Σε μια τέτοιου είδου συνεδρίαση συνήθως έχουμε την ε, ψυχρότητα των ε, αριθμών και το βάθος ε, του ανθρώπινου δράματος από την άλλη. Ακούσαμε πρώτα το ανθρώπινο δράμα και θα ήθελα ωστόσο αυτή τη στιγμή να σας θυμίσω κάποια στοιχεία αλλά και κάποιες αρχές. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι η λύση στην κρίση. Είναι η συνέπεια της κρίσης. Είναι η συνέπεια, ε, επαναλαμβάνω, της κρίσης και όχι η λύση η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ανεξάρτητη, ουδέτερη και αμερόληπτη. Αυτές είναι οι βασικές αρχές επί των οποίων ε, βασίζεται, ε, δράζεται εδώ και δεκαετίες και τις οποίες αρχές έχει ε, υιοθετήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακριβώς η έλλειψη πολιτικής λύσεως στην κρίση αυτή καθιστά σήμερα λόγω του είδους της σύγκρουσης όπως θύμισε και ο συνάδελφος ε, την οποία αντιμετωπίζουμε που καθιστά την ανθρωπιστική βοήθεια καθημερινά πιο δύσκολη. Η πραγματικότητα λοιπόν που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι εξή. Σήμερα εκτιμάμε τον, αριθμό των ε, θυμάτων ε, στις 100.000 ανθρώπους περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι Σύριοι εντός της επικράτειας της Συρίας χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια και από αυτά τα 7 εκατομμύρια άνθρωπους περίπου τα 4 είναι εκτοπισμένα εντός της επικράτειας της Συρίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UNICEF, όπως έλεγε ο συνάδελφος, περίπου 50% αυτού του πληθυσμού αποτελείται από παιδιά μικρής ηλικίας και από νέους. Όσον αφορά τις γειτονικέ χώρες, α, ναι, να πω και δύο λόγια για ε, έναν πληθυσμό που έχει καταστεί ιδιαίτερα ευάλωτος λόγω αυτής της κρίσης που είναι οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες που ήταν εγκατεστημένοι στη Συρία. Από τους οποίους το 80% αυτή τη στιγμή χρειάζεται ε, ανθρωπιστική βοήθεια είτε εντός της Συρίας είτε στις γειτονικές χώρες όπου έγιναν δεκτοί μετά από ε, διαδοχικές μετακινήσεις. Όσον αφορά τον αριθμό των προσφύγων, εκτιμά το αριθμός τους σε 1.700.000 άνθρωποι. 560.000 στο Λίβανο, 500.000 στην Ιορδανία και στην Τουρκία έχουμε φτάσει σήμερα περίπου τις 400.000 πρόσφυγες. Αλλά βέβαια οι ε, εκτιμήσεις αυτές θα πρέπει να τελειοποιηθούν. Ε, τώρα, ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν ε, οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια ή καταρχήν πρόσβαση στη Συρία. Από τη μια πλευρά η κυβερνητικές αρχές πολλαπλασιάζουν τα γραφειοκρατικά και διοικητικά εμπόδια για την δρομολόγηση του, της ανθρωπιστικής βοήθειας και από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση, η αντίσταση είναι πολύ κατακαιρματισμένη σε βαθμό που χρειάζεται ώρα με την ώρα και λεπτό με το λεπτό να διαπραγματεύεται κανείς ε, το πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να φτάσει σε όλες τα ε, άκρες της χώρας, ε, σε όλη την επικράτεια. Είτε είναι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης σε τα συγκεκριμένα μέρη είτε όχι. Στις γειτονικέ χώρες, προφανώς ο Λίβανος έχει φτάσει σήμερα, μάλλον έχει ξεπεράσει το όριο ε, απορρόφησης όλου αυτού του κόσμου και η Ορδανία παρατηρούμε και η κυρία Γεωργίευα μόλις ε, στις αρχές της εβδομάδας πήγε εκεί ε, παρατηρείται ένα φαινόμενο αυξανόμενο εντάσεων για απόλυτα ανθρώπινους λόγους εντάσεων ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους και τις κοινότητες υποδοχής. Νομίζω πως όλοι πρέπει να χαιρετήσουμε την εξαίρετη προσπάθεια υποδοχής που γίνεται και στηρίζεται αυτή τη στιγμή από τις γειτονικέ χώρες, τις δυο που ανέφερα, αλλά και την Τουρκία, αλλά και σε ένα μικρότερο βαθμό, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε, το Ιράκ. Από ανθρωπιστικής άποψης προφανώς η κατάσταση θα πρέπει να εξεταστεί λοιπόν σε μια προοπτική που βασικά είναι μια προοπτική περιφερειακή. Το να αντιμετωπίσει κανείς μια ανθρωπιστική καταστροφή τέτοιο εύρους ε, απαιτεί την κινητοποίηση μέσων άνευ προηγουμένου. Γενικά νούμερα αναφέρθηκαν από το συνάδελφο πριν από λίγο, ενώ όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια αυστηρά, είχα την ευκαιρία να το θυμίσω σε άλλη επιτροπή του Κοινοβουλίου αυτού πριν από δύο μέρες, έχουμε χρησιμοποιήσει το φθινόπερο μισό δις ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Συρία 50% περίπου αυτού του ποσού, η Ορδανία και Λίβανο. Δεσμεύσαμε δηλαδή 500 εκατομμύρια το φθινόπωρο. Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία. Και εδώ αυτά τα λέω από τον έλεγχο του κ. Οκτάη που είναι ο υπεύθυνο τη τουρκική κυβέρνηση, με την οποία είχαμε μια εξαίρετη συνεργασία στη διάρκεια τούτης εδώ της εβδομάδας. Όπως έλεγα, η προσπάθεια υποδοχής που γίνεται από την κυβέρνηση της Τουρκίας στηρίζεται, όπως είπα, από την κυβέρνηση, από τους δικούς της πόρους. Είναι πραγματικά θεαματική και σημαντική η προσπάθεια αυτή. Αυτή τη στιγμή περίπου 200.000 πρόσφυγες φιλοξενούνται σε καμιά εικοσαριά καταβλισμούς σε δέκα επαρχίες και τρεις άλλες εγκαταστάσεις υποδοχής κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή. Είναι ένα φαινόμενο που φαντάζομαι και ο Σοκτάι θα το αναφέρει περισσότερο, ένα φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερο η Τουρκία σήμερα είναι οι πρόσφυγες εκτός των καταβλισμών, δηλαδή στις αστικές περιοχές, των οποίων ο αριθμός είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, γιατί δεν είναι όλοι καταγεγραμμένοι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ανθρωπιστικών οργανώσεων, και των διεθνών ε, υπηρεσιών του ΟΗΕ, όπως είπατε η αρμοστία, πρόκειται για 300 με 400 χιλιάδες σήμερα Οι αναλογίες αυτές είναι δραματικές για την Τουρκία. Αλλά τι δεν είναι δραματικό σε μια τέτοια κατάσταση. Μια λογική εκτίμηση θα ήταν ότι η Τουρκία θα χρειαστεί να υποδεχτεί μέχρι το τέλος του έτους ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Συρία. Να πω ότι έχουμε μετρήσει τις δραματικές συνέπειες της μάχης γύρω από το Κούσα, ενώ ετοιμάζεται μια μεγάλη μάχη γύρω από το Χαλέπι, που είναι μια μεγάλη πόλη περίπου 4 εκατομμυρίων ανθρώπων υπό κανονικές συνθήκες. Είναι σαφές ότι θα έχουμε ακόμα ένα παράγοντα επιδείνωσης πέρα από τα όσα είχαμε φανταστεί μέχρι τώρα όσον αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση. Συνεργαστήκαμε λοιπόν με την Τουρκία με διάφορα χρηματοδοτικά μέσα μέχρι στιγμής το συνολικό ποσό συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία έχει ανέλθει σε ένα σχετικά μικρό ποσό. Σχετικά μικρό ποσό πρέπει να το πούμε. Είμαστε περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Η συνεργασία λοιπόν ανθρωπιστικής βοήθειας και ο κ. Σουκτέι το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ε, επηρεάζεται από το είδος της ανθρωπιστικής πολιτικής που είχε η τουρκική κυβέρνηση που ήταν ε, κατευθυνόμενη από τις, από τις δημόσιες αρχές. Η υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης που αντιπροσωπεύω σήμερα εδώ και η κυρία Γεωργίευα εργάζονται με βάση την εντολή τους με οργανώσεις υπηρεσίες των, των, του ΟΗΕ, και μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Συνεργαστήκαμε με την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες σε δράσεις που διοργάνωσε η ίδια σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του κυρίου Οκτάη, αλλά κυρίως χρησιμοποίησαμε άλλα μέσα και όχι αυτά τη ανθρωπιστική βοήθεια, για να βοηθήσουμε την ΦΑΝΤ στην προσπάθεια υποδοχής και στην οικοδόμηση των απαραίτητων μέσων για να υποδεχτεί, όπως είπαμε, τους πρόσφυγες. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουμε και η, κυρία, η επίσκεψη του κυρίου Κτέη μας προετοίμασε γι' αυτό. Θα περάσουμε σε μια ε, μεγαλύτερη ταχύτητα όσον αφορά την τεχνική και οικονομική βοήθεια με τους ε, Τούρκους και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, τις τουρκικές που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Έχουμε διερευνήσει διάφορους οδούς συνεργασίας που κυρίως αφορούν την υποδοχή και την κάλυψη των αναγκών, των ιατρικών αναγκών αυτού του πληθυσμού που όπως είπα πριν από λίγο είναι οι, αστι... οι πρόσφυγες στα αστικά κέντρα. Θα έλεγα όμως ότι στην Τουρκία όπως και αλλού βρισκόμαστε μόνο στις αρχές της συνειδητοποίησης και της αντιμετώπισης ε, ε, των ανθρωπιστικών ε, συνεπειών αυτής της πολιτικής και ανθρώπινης καταστροφής που αντιπροσωπεύει η κρίση στη Συρία. Η κατάσταση είναι πολύ οξυμένη, παίρνει διαστάσεις άνευ προηγουμένου και από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να πάψει για την ώρα. Και επειδή αναφέραμε και θα αναφέρουμε και στη σημερινή συζήτηση την προοπτική, μάλλον την έλλειψη προοπτικών για πολιτική λύση, ε, όμως είναι προφανές ότι ακόμα και αν βρεθεί πολιτική λύση στους επόμενους μήνες, ποιος ξέρει, το επίπεδο της καταστροφής στην Συρία και στην περιφέρεια αυτή είναι τέτοιο που οι ανθρωπιστικές συνέπειες της σύγκρουσης που ζούμε σήμερα θα διαρκέσουν και θα επιβαρύνουν τις γειτονικές χώρες για πολλά χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τιμπρόε. Ακόμα και αν ε, έχουμε αυτή την ενοχλητική τάση να συνεχίζουμε αυτές τις προσπάθειες που είναι αυτοεκπληρούμενες. Δηλαδή προβλέπουμε για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, αλλά αυτή η προοπτική ότι ε, θα προετοιμαστούμε για ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, αυτό σημαίνει πόσοι νεκροί ακόμα και πόσες χιλιάδες ε, και πόσα θύματα αυτά. Είναι αφόρητη η προοπτική και ενδεχομένω μια ε, πολιτική πρωτοβουλία χρειάζεται. Επιτέλους κάποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι πρόθυμες να υποστηρίξουν και στρατιωτικά ε, την αντιπολιτευτική. Θα ήταν ενδιαφέρον, κύριε Χατύπ, δεν αναφερθήκατε ιδιαίτερα σε αυτό, να δούμε ε, πώς μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί ενδεχομένως να αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και πολιτικό. Διότι, όπως είπατε, η στρατηγική της ε, κυβέρνησης του καθεστώτος είναι να κερδίζει χρόνο και μέχρι τώρα μάλλον τα έχει καταφέρει και ενδεχομένως αυτή η πρωτοβουλία της ΝΕΒΙΣ 2 που αν κατάλαβα καλά ε, υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το γνωρίζω, ε, συνεχώς αναβάλλεται μέρα με τη μέρα και εβδομάδα με τη εβδομάδα. Και αυτό είναι παρακιστική τακτική και στρατηγική που κάνει τον Άσαντ να κερδίζει χρόνο. Νομίζω πρέπει να βρούμε κάποια άλλη προοπτική αυτό παρά να ε, παίζουμε τις καθυστερήσεις μήνα με το μήνα να παρατείνουμε αυτό το τρόμο και τη φρίκη που είναι γνωστή. Ε, θα συνεχίσει ο κύριος Οκτάη και χαίρομαι που μαθαίνω ότι έχετε συντονίσει και τελειοποιήσει τα θέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεδομένης της ε, παρουσίας σας εδώ και έχετε μια ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια προσφύγων. Όπω πολλοί συνάδελφοι έχω επισκεφθεί εγώ αυτούς του καταβλισμού. Είναι πολύ εντυπωσιακή η δράση, ε, πολύ αποτελεσματική και είναι και κρατική. Όπως είπατε δεν ε, ε, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρήκατε όμως άλλους τρόπους να τα ε, ρυθμίσετε για να σας υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι πολύ μεγάλη και η χρηματική σας επιβάρυνση. Ο κύριος Οκτάη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη συμπρόεδρη της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί βουλευτές, κύριε Χετύπ, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που εντάξατε στην ημερήσια διάταξή σας ένα τόσο σημαντικό θέμα. Εμείς πράγματι ως Τουρκία κάνουμε πολλά προς την κατεύθυνση αυτή και έχουμε τώρα την ευκαιρία να συμμεριστούμε μαζί σας τις σκέψεις μας και να σας ενημερώσουμε. Ε, είναι πολύ σημαντικά βέβαια αυτά που κάνουμε εμείς, αλλά ακούγοντας τον κύριο Χατίμπ, για την αίσθηση ότι είναι μια τρύπα στο νερό περίπου όλα αυτά που κάνουμε. Διότι ό,τι και να κάνουμε, όλες μας τις προσπάθειες για να ε, αναπτύξουμε, η λύση δεν ε, θα έρθει στο αμυγός ανθρωπιστικό επίπεδο. Η λύση πρέπει να είναι σε πιο πολιτική βάση μέχρι να βρεθεί μια πραγματική λύση απέναντι σε αυτό το δράμα, απέναντι σε αυτά τα δεινά και το θρήνο του λαού στη Συρία. Θα πρέπει να περιορίσουμε στο ελάχιστο ε, ε, αυτή τη ε, κατάσταση, τη τραγωδία και να είμαστε στο πλευρό τους. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χατύπ και τους υπολείπους συμμετέχοντες. Ευχαριστώ για την παρουσίαση της κατάστασης στη Συρία και την ανθρωπιστική και αν μου επιτρέπετε θα σας μιλήσω εγώ για πιο τεχνικά στοιχεία, να σας εξηγήσω τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τι χρειαζόμαστε στο προσεχές μέλλον και πώς μπορεί να βοηθήσει η διεθνής κοινότητα για να αναλάβει και τις δικές της ευθύνες. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν θα σας εκθέσω την κατάσταση. Στις 22 Απριλίου του 2011 η Τουρκία de facto έγινε μέρος ε, αυτού του θέματος ε, από την ανθρωπιστική σκοπιά βέβαια. Οι πρώτοι που έφτασαν από το Χατάι του Μπεγκεζού ήταν 252. Περίπου μόλις ξέσπασε η κρίση. Άνοιξε αμέσως τα σύνορά της η Τουρκία και δήλωσε ότι δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηρή απέναντι σε αυτό το ανθρωπιστικό δράμα. Ξέρετε, δεν ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε αυτό. Το έχουμε ξανακάνει για τη Βοσνία, για τη Βουλγαρία, για το Ιράκ, ε, για τη Βυρμανία, Μιανμάρ δεχόμαστε ε, πρόσφυγες και σήμερα δείχνουμε την ίδια ευαισθησία απέναντι στη Σύρια σε ό,τι αφορά ε, τώρα θέματα ε, θρησκείας, φίλου, φίλης δεν μας απασχολούν. Όποιος έρχεται στην Τουρκία και ζητάει βοήθεια του τη δίνουμε. Στις 29 Απριλίου λοιπόν του 2011 άρχισε αυτή η προσπάθεια γύρω ε, στο Χατάι στην Αντιόχεια ήταν 252 μικρός ο καταβλισμός πρώτα 3-4 χιλιάδων ακολούθησε ένας δεύτερος και ένας τρίτος και ένας τέταρτος γιατί δεν χωρούσαν πλέον οι πρόσφυγες. Ε, επίσης, ε, ε, στη συνέχεια χάλασε ο καιρός. Ερχόταν ο χειμώνας και η κυβέρνησή μας μετά από εντολή του Πρωθυπουργού έκανε και νέους καταβλισμούς για να αντιμετωπίσει το χειμώνα γιατί φαινόταν ότι η κατάσταση αυτή δεν ήταν καθόλου προσωρινή. Αρχίσαμε λοιπόν να χτίζουμε περίπου πόλεις ε, με κοντέινερ ε, στους καταβλισμούς στην πόλη του Κιλής και μάλιστα ε, τις χαρακτηρίζουμε έτσι πόλεις σε κοντέινερ και όχι καταβλισμούς, όχι στρατόπεδα, διότι δεν πρόκειται για καταβλισμούς, δεν είναι σκηνές. Είναι πραγματικά κοντέινερ, είναι πιο γερές κατασκευές για να περάσουν το χειμώνα. Και επίσης θέλαμε να δώσουμε την αίσθηση στον κόσμο ότι ζει σε πόλη. Σε ό,τι αφορά τώρα το νομικό καθεστώς, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί ε, έχουν ένα καθεστώς προσωρινής προστασίας και τους ονομάζουμε φιλοξενούμενους, προσκεκλημένους μας. Δεν θέλουμε να τους ε, χαρακτηρίσουμε πρόσφυγες οι άνθρωποι που χρειάζονται προσωρινή διεθνή προστασία. Θέλουμε να τους δείξουμε ότι τους φιλοξενούμε στην Τουρκία, να καταλάβουν την τουρκική φιλοξενία και να αισθανθούν ότι είναι προσκεκλημένοι μας, γιατί τους καλέσαμε. Ε, και θέλουμε να τους ε, δεχτούμε στη χώρα μας, στο σπίτι μας. Σε αυτές λοιπόν τις πόλεις τα κοντέινερ ήταν σημαντικό να γνωρίζουν και οι εργαζόμενοι ότι υποδέχονται προσκεκλημένους, καλεσμένους και έτσι θα πρέπει να τους φέρονται. Ότι είναι σαν να φιλοξενείς κάποιον στο σπίτι σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εκατέρωθεν αντίληψη της κατάστασης. Εκεί λοιπόν αυτή η πόλη κοντέινερ που ήταν και μάλιστα ε, ε, πολύ πιο ψηλά από τα διεθνή πρότυπα ε, μπόρεσαν να φιλοξενηθούν 10.000 αλλά ούτε αυτό έφτανε, διότι η κατάσταση συνεχιζόταν επιδεινούμενη στην Τουρκία και στο Αντέπ, κοντά στο Γκαζί Αντέπ, επίσης ε, φτιάξαμε ένα νέο καταβλισμό, Ισλάριε, και πάλι δεν έφτασε αυτό και πήγαμε σε άλλες πόλεις και σήμερα είναι περίπου 10 οι καταβλισμοί αυτοί που είναι πόλεις με, ε, με κοντέινερ 10 και 21 καταβλισμοί με σκηνές. και έχει περίπου καλυφθεί η δυνατότητα υποδοχής, είναι 100% δηλαδή. Το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού και η πολιτική προστασία, η υπηρεσία θεομηνιών έχει επιληφθεί αυτής της προσπάθειας και πάντα στα πλαίσια των εργασιών μας προσπαθούμε να τα ε, διοργανώνουμε. Και πάλι ε, πρέπει να σας πω ότι υιοθετήσαμε την εξής αρχή. Ε, Βεβαίω υπάρχει μια ανθρωπιστική διάσταση, αλλά εμεί δεν θέλουμε μια λύση ε, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άπαξ. Διότι ε, ο κόσμος δεν ζει σε συνθήκες έτσι προσωρινής διαβίωσης. Είναι μια μόνιμη, μονιμότερη κατάσταση. Ας πούμε, όταν κάποιος είναι άστεγος, Μπορεί για μία μέρα να τον φιλοξενήσεις σε ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων ή να τον καλέσει σε ένα πολύ ακριβό εστιατόριο, αλλά την άλλη μέρα πάλι άστεγος θα είναι. Γι' αυτό εμείς δεν θέλαμε προσωρινές λύσεις και μεσοβέζικες, δεν θέλαμε καταβλισμού με σκηνέ, δεν θέλαμε ε, ε, πόλεις, με κοντέινερ, με υγειονομικέ υπηρεσίε, με σχολεία. Ε, έχουμε επίσης και ε, επιμελητεία ε, για την παροχή τροφίμων, άλλων εφοδίων ε, πέρα από τρόφιμα, με κέντρα διαχείρισης ε, και όταν μιλούμε για υγειονομική περίθαλψη, πρόκειται για 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε επίπεδο πολυκλινικής και πάνω από 200.000 είναι εκείνοι που αυτή τη στιγμή ε, εποφελούνται από τις υπηρεσίες υγείας. Και όταν δεν αρκεί αυτό ε, μπορούν να μεταβούν στα νοσοκομεία της περιοχής. Και πάνω από 15.000 έχουν ήδη χειρουργηθεί. Πάνω από 24.000 είναι ε, αισθενείς που νοσηλεύονται. Πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας έχουμε αυτή την πρόβλεψη επίσης για τις υπηρεσίες υγείας. Στη συνέχεια καλέσαμε και το Υπουργείο Υγείας να αναλάβει εκείνο την περίθαλψη και όχι πλέον η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Θεομηνιών. Με τον ίδιο τρόπο απευθυνθήκαμε και στο Υπουργείο Παιδείας για να μπορούν τα παιδιά να ζήσουν μια φυσιολογική όσο γίνεται ζωή. 30.000 παιδιά περίπου πηγαίνουν σχολείο από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τελευταία τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ορισμένοι μπορούν μέχρι και πανεπιστημιακά μαθήματα να παρακολουθούν με την αρμόδια υπηρεσία για την ανώτατη παιδεία, η συνεργασία. Επίσης έχουμε επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ε, ενηλίκων για να μπορούν να εκπαιδεύονται και να παρακολουθούν μαθήματα, ε, είτε είναι υπολογιστές, πληροφορική, κοπτική, ραπτική. Είναι 300 περίπου τα μαθήματα που μπορούν να επιλέγουν οι ενήλικες και χιλιάδες έχουν λάβει και πιστοποιητικά και ενδεικτικά ε, εκπαίδευση ενηλίκων. Εκεί έχει επιφορτιστεί με αυτό το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Ε, βεβαίως συντονιζόμαστε μαζί τους, αλλά το έχουν αναλάβει εκείνοι. Και σε ό,τι αφορά ε, το περιεχόμενο, το πρόγραμμα σπουδών, αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, ε, ε, σε πολύ αγαστή συνεργασία λοιπόν μαζί μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τον επισητισμό, συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Γεωργίας η ασφάλεια ε, εξαρτάται από το Υπουργείο Εξωτερικών κτλ. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια δεν είναι μόνο στους δικούς μας ώμους, κάθε Υπουργείο να λαμβάνει τις ευθύνες του στον τομέα του. Στους καταβλισμούς αυτούς λειτουργεί καλά αυτή η προσπάθεια. Είναι ένα σύστημα πάρα πολύ ε, καλό, υγιές και εύρωστο και διαρκεί εδώ και δύο χρόνια. Και τελικά ε, είτε καταβλισμό ονομάζει ένα τέτοιο σχηματισμό, είτε πόλη, τελικά καταβλισμό είναι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανεί να βγει και είναι εκεί μέσα κλεισμένο, τελικά γίνεται φυλακή. Και εμεί δεν θέλαμε τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό εδώ και δύο χρόνια προσπαθούμε να διοργανώσουμε καλέ υπηρεσίε στου καταβλισμού αυτού, αλλά όσο καλέ και να είναι υπηρεσίε, ο καταβλισμό παραμένει στρατόπεδο. Ε, και κάποια στιγμή ε, γνωρίζει και τα όρια του ως προς τη δυνατότητα υποδοχής. Η τραγωδία συνεχίζεται και επίσης είχαμε και σύρους που δεν επιθυμούσαν να ενταχθούν σε ένα τέτοιο καταβλισμό. Όσο σύγχρονες εγκαταστάσεις και να είχαν, εκείνοι επιθυμούσαν ενδεχομένω να παραμείνουν σε πόλεις, να νοικιάσουν ένα σπίτι όταν είχαν την ευκαιρία να το κάνουν. Μετά από ένα χρόνο όμως ή κάποιο διάστημα που δεν είχαν πλέον οικονομικούς πόρους, υποχρεώθηκαν και αυτοί να έρθουν στους καταβλισμούς. Ε, επίσης είχαμε κάποιους πρόσφυγες που δεν πέρασαν τα σύνορα με τρόπο νόμιμο, με διαβατήριο, αλλά όταν ήταν μαζικοί οι βομβαρδισμοί ε, ήρθαν από άλλες οδούς. Πάνω από 300.000. Σήμερα έχουμε πάνω από 500.000, μισό εκατομμύριο Σύρους δηλαδή στην Τουρκία. Στην αρχή εμείς επικεντρωθήκαμε εκεί στους καταβλισμούς, αλλά μετά αρχίσαν τα προβλήματα εκτός των καταβλισμών. Και πώς θα αντιμετωπίσεις τα προβλήματα των ανθρώπων αυτών που είναι αλλού. Εκεί και πάλι ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, προσπαθήσαμε να τους παρέχουμε στην αρχή υπηρεσίες υγείας και τώρα ε, μπορούν, όπως κάθε Τούρκος πολίτης, να απευθύνονται στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή όμως έχουν εγγραφεί σε κάποιο μητρό ως ΣΥΡΙ πρόσφυγες. Και από εκεί και πέρα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Ε, αλλά αυτό όμως έχει επιβαρύνει τώρα τα νοσοκομεία ε, στις παραμεθόριες πόλεις μας και τις δομές υγείας και εκεί προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να αυξήσουμε τις δυνατότητες υποδοχής. Ε, ήταν τέτοια η αύξηση του πληθυσμού και των αριθμών που εμφανίστηκαν και νέες ανάγκες και προσπαθούμε να ε, βρούμε μια πιο συστηματική λύση απέναντι σε αυτές. Είτε πρόκειται σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους διεθνείς οργανισμούς. Ανέκαθεν λοιπόν το θέτουμε υπόψη σε αυτό. Έχουμε φτιάξει αυτό το σύστημα που λειτουργεί και είπαμε ότι έχουμε ένα σύστημα που λειτουργεί καλά στους καταβλισμούς που έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του και μπορούμε ε, να το κάνουμε και εκτός των καταβλισμών. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε χώρο. Βλέπετε εδώ μερικές φωτογραφίες ακόμα για τους καταβλισμούς. Ε, θα πρέπει να χτιστεί ένα τέτοιο σύστημα για να μπορέσουμε να καταγράφουμε όλους αυτούς τους πρόσφυγες που επαναλαμβάνω θεωρούμε εμείς φιλοξενουμένους, προσκεκλημένους μας, guests και ε, οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν να κάνουν μια αξιολόγηση των αναγκών, ε, μια εκτίμηση των αναγκών για να μπορέσουμε να δούμε τι χρειάζεται και να καλύψουμε τις ανάγκες. Ε, από τη στιγμή που έχει εγγραφεί κάποιος ένα μητρό, μπορείς να πεις ότι έχει τις τάδε ανάγκες ε, περίθαλψης ή τις δίνει ανάγκες εκπαίδευσης ή ε, επισητισμού. Ε, αλλά θα πρέπει να τους γνωρίζουμε. Έχει αρχίσει αυτή τη διαδικασία. Σήμερα είναι πάνω από 70.000 οι Σύριοι που βρίσκονται εκτός των καταβλισμών σε διάφορες πόλεις, έχουν έρθει να εγγραφούν στο σύστημα και τέλος Αυγούστου θα αρχίσει να επεκτείνεται ε, αυτή η προσπάθεια και εκτός των καταβλισμών. Και θα έχουμε και βιομετρική καταγραφή που θα λειτουργήσει ακόμα καλύτερα και θα είναι ακόμα πιο ε, ασφαλής. Αλλά αυτά δεν μας αρκούν. Βλέπουμε αυτή ποια είναι η ζήτηση τώρα. Όταν έρχεται κάποιος να εγγραφεί γνωρίζουμε τι ζήτηση υπάρχει. Αλλά επίσης θα πρέπει ε, να καταγράφονται και οι δωρητές και η προσφορά, όχι μόνο η ζήτηση. Δηλαδή ποιο παρέχει πιο εξοπλισμό. Ε, και θα τους δώσουμε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό για να μπορούν να εγγράφονται στο σύστημα και online ε, μπορεί κανείς αμέσως να βλέπει ποιος δίνει ποια ε, βοήθεια και ποιες είναι οι ανάγκες. Και θα μπορεί ο καθένας να δεσμεύεται ότι εγώ μπορώ να δωρήσω ή να δώσω το τάδε. Και αμέσως βλέπουμε τις υποσχέσεις δωρεών έτσι ώστε με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο να μπορούμε στη συνέχεια να δίνουμε ε, αυτές τις δωρεές στους δικαιούχους. Έχουμε αρχίσει να φτιάχνουμε το λογισμικό για το σύστημα αυτό και εδώ και δύο μήνες λειτουργεί. Στην πρώτη φάση είχαμε το εξής πρόβλημα σε σχέση με τη διεθνή κοινότητα. Πολλοί έλεγαν ότι θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά να πάμε στους καταβλισμούς για να βοηθήσουμε επιτόπου. Και αν ξέραμε τις ανάγκες, αν μπορούσαμε επιτόπου να δούμε τι χρειάζεστε, θα σας βοηθούσαμε. Και εμείς ανέκαθεν λέγαμε και πιέζαμε ότι, κοιτάξτε, η ΜΚΟ είναι χιλιάδες. Δεν μπορούμε να αφήνουμε κάθε μη κυβερνητική οργάνωση να μπαίνει στους καταβλισμούς. Αλλιώς θα πρέπει να χρειάζεται να διαχειριζόμαστε τους μη κυβερνητικού οργανισμούς, αντί να διαχειριζόμαστε τη βοήθεια. Και τους είπαμε, εγγραφείτε, υπάρχει το σύστημα ηλεκτρονικά. Βέβαια σε μια δεύτερη φάση τους είπαμε ότι είναι ελεύθερη η πρόσβαση στον καταβλισμό από τη στιγμή που θα έχετε εγγραφεί όμως το σύστημα. Ε, και εκεί πηγαίνετε επί τόπου και αν θέλετε να διαχειριστείτε τη βοήθεια που παρέχετε οι ίδιοι. Και ξαφνικά όλες αυτές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που είχαν τέτοια λαχτάρα να πάνε στους καταβλισμούς, ε, ε, πολύ λίγες ήταν αυτές που εμφανίστηκαν επί τόπου για να βοηθήσουν, πέντε τον αριθμό. Κανένας άλλος δεν έδωσε σοβαρή απάντηση και υπόσχεση δωρεάς. Ποιο είναι το κόστος ε, όλων αυτών των προσπαθειών για την Τουρκία. 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Και όχι μόνο στο εσωτερικό της Τουρκίας. Πολλοί άλλοι θέλησαν να μεταβούν στη Συρία, αλλά τελικά δεν το έπραξαν. Και 150 εκατομμύρια δολάρια ε, πήγαν στη Συρία με νόμιμο τρόπο δια των ε, διάβλων των Ηνωμένων Εθνών. Ε, σε ό,τι αφορά την εξωτερική βοήθεια, η συνολική εξωτερική βοήθεια που έλαβε η Τουρκία μέχρι σήμερα ήταν 107 εκατομμύρια δολάρια μόλις. 107. 50 εκατομμύρια σε ρευστό από την ε, Σαουδική Αραβία, 36 εκατομμύρια δολάρια από τα Ηνωμένα Έθνη, το ύπατη αρμοστία συγκεκριμένα, και ε, από άλλους οργανισμούς που συνδέονται με τα Ηνωμένα Έθνη. Και είχαμε και, ε, αυτά είναι ηλική βοήθεια, όχι σε χρήμα, σε εξοπλισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της δηλαδή, έχουν δώσει κάποια βοήθεια ως κράτη. Να σας δώσω μερικούς αριθμούς. 26.000 η Αυστρία, 145.000 δολάρια η Γαλλία, χιλιάδες. Ο Γερμανικός ε, Ερυθρός Σταυρός 135.000, η ε, Σουηδία 20.000, η Ολλανδία 2,5 εκατομμύρια, το Βέλγιο για να χτιστεί ένα σχολείο 650.000 ευρώ. Ιδού το σύνολο της βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Μπάουερ είπε προηγουμένως κάτι για 30 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί συμπεριλαμβάνεται και τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών. Εγώ δεν ξέρω, τα δικά μας αριθμητικά στοιχεία αυτά λέγουν. Και σε ό,τι αφορά τον ΟΗΕ, ε, πάνω, ε, περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια ε, θα μεταφερθούν στη χώρα και να σας δώσω μερικά στοιχεία ακόμα, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά τη δράση επιτόπου. 4,2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα καλύπτονται από σκηνές στους καταβλισμούς. Και όταν φτάσαμε στο 1 εκατομμύριο τετραγωνικά, από εκεί και πέρα χρειάζονται και κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή, είναι 17 ε, Συνολικά 8 εκατομμύρια τετραγωνικά ε, σε πόλεις κοντέινερ, 145.000 ε, σκηνές χρειαζόμαστε περαιτέρω, πέρα από τις σκηνές που έχουμε, που είναι τώρα 30.000 και 10.000 τα κοντέινερ. Όταν φτάσουμε λοιπόν στο 1 εκατομμύριο τετραγωνικά, η κατάσταση γίνεται δύσκολη. Και ιδίω εκεί, σε αυτή την πλατφόρμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, και, αλλά και τις χώρες μεμονωμένα, είτε μεμονωμένα είτε ως Ένωση, πρέπει πραγματικά να εγγράψετε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Εμείς ως Τουρκία έχουμε κάνει να λειτουργεί πραγματικά το σύστημα. Τα Ηνωμένα Έθνη άλλωστε το παραδέχονται. Και η Ένωση επίσης. Μας λένε τόσο καλά τα καταφέρνετε που μπορείτε να το κάνετε, να τα αφήσουμε σε εσάς. και φαίνεται σαν να έχουν την εντύπωση ότι δεν έχουμε ανάγκη από τίποτε. Εμείς ως Τουρκία δεν ζητούμε βοήθεια, εμείς ζητούμε στήριξη γιατί είναι ένα πρόβλημα περιφερειακό, δηλαδή είναι στην περιφέρειά μας, ο καθένας βεβαίως πρέπει να αναλάβει τις ευθύνε του και ε, να, στήριξη, να υπάρξει στήριξη. Αυτά που κάνει η Τουρκία και αυτά που γίνονται για την Συρία ε, πρέπει να δείξουν και κάποια ευαισθησία. Αυτό ζητούμε. Μιλήσαμε για πολιτική ανοιχτών θυρών, την οποία εφαρμόσαμε. Αλλά βεβαίω και υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχει και η ανθρωπιστική διάσταση. Ακούμε καμιά φορά ότι η Τουρκία επιβραδύνει τις εισόδους στις, ε, στα σύνορά της δεν επιτρέπει σε όλους πρόσφυγες να εισέρχονται. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω. Ορισμένες οργανώσεις που ισχυρίζονται ότι ανοίγουμε και κλείνουμε τα σύνορά μας, διεθνείς οργανώσεις ή και χώρες, δεν έχει τόση σημασία, αυτοί ή αυτές έχουν δεχθεί πρόσφυγες. Κάθονται στο θεωρείο και παρακολουθούν τα τεκτενόμενα χωρίς να συμμετέχουν. Είναι απλοί θεατές. Ενώ όλοι πρέπει να ρηχτούμε στην δουλειά. Και, όλοι και όλες οι χώρες δηλαδή πρέπει να ασκήσουν αυτή την πολιτική των ανοιχτών θυρών. Ναι, ακούμε από τις χώρες αυτές ότι α, και αυτές ανοίγουν τα σύνορά τους. Τι είναι τώρα τα σύνορα της Τουρκίας ή της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Ενωμένου Βασιλείου, του Βελγίου. Βεβαίως, μπορούμε να βάλουμε και πτήσεις. Να βάλουμε τους ανθρώπους αυτούς σε αεροπλάνα και να τους στείλουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εάν και αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες θελήσουν να ασκήσουν την πολιτική των ανοιχτών θυρών. Άλλο θέμα. Εάν φτάσουν οι πρόσφυγες στο ένα εκατομμύριο, αυτά όλα που κάνουμε δεν θα αρκέσουν. Θα πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Ίσως μια buffer zone ή μια ζώνη προστασίας, ίσως κάποια άλλη πολιτική θα πρέπει να εκπονηθούν άλλες λύσεις. Το σύστημα που σας εξήγησα προηγουμένως, όπου μας έλεγαν οι διάφορες μη κρατικέ οργανώσεις «Α, αφήστε μας να μπούμε στους καταβλισμούς» και τα λοιπά και τελικά δεν ήρθαν. Βεβαίω υπάρχουν προβλήματα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των καταβλισμών και σε αυτά μπορούν να συμβάνουν μπορούν να ε, κάνουν δωρεές υλικές σε είδος, μπορούν να φτιάξουν σχολεία, μπορούν να προσφέρουν ε, επισητιστική βοήθεια, ό,τι θέλετε. Έχουμε συγκεκριμένα ε, σχέδια, σοβαρά, project, όποιος θέλει μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά. Θέλω σιγά σιγά να καταλήξω, τονίζοντας και πάλι ότι οι λύσει που θα πρέπει να δοθεί θα πρέπει να είναι πολιτική. Και το πρόβλημα της Συρίας θα πρέπει να λυθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα με ειρηνικό τρόπο μέσα στην ίδια τη Συρία ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να επιστρέψουν στις αιστείες τους. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφραστώ. Ο Συμπρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, λεπτομερείς αυτές εξηγήσεις που δώσατε. Επανέρχομαι σε κάτι που είπατε. Η ανθρωπιστική βοήθεια που πρέπει να δοθεί, όντως πρέπει να δοθεί. Το γεγονός ότι υποδέχεστε, υποδεχόμαστε δηλαδή τους εκτοπισμένους ως αδελφούς, βεβαίως και θα φροντίσουμε τις ανάγκες τους. Αυτό για μας είναι αυτονόητο. Αλλά δεν αρκεί. Δεν πρόκειται μοναχά για μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν σωστά οι ανάγκες των προσφύγων. Πρέπει να καταπολεμηθεί το πρόβλημα, να λυπηθεί το πρόβλημα στη ρίζα του. Και αυτό είναι δείγμα ανθρωπιάς, γιατί οι άνθρωποι είναι. Ανθρώπινες ζωές. Και αυτές πρέπει να διαφυλάξουμε. Όχι λοιπόν μόνο να φροντίσουμε τους πρόσφυγες, πρέπει να τεθεί ενώπιον των ευθυνών του το ίδιο το Συριακό καθεστώς. Η Τουρκία βέβαια έχει ιδιαίτερο ρόλο να παίξει, όπως εξηγήσατε. Αλλά ρόλο έχει να παίξει και η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της. Βέβαια, τα Ενωμένα Εθνή και άλλοι φορείς είπαν ότι η Τουρκία τα καταφέρνει καλά. Όμως, όπως εξήγησε ο κ. Σοκτάι, παρόλα αυτά, δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει δυνατότητα το συντομότερο δυνατό οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν Ναι, λέει η κυρία Φρότ, βεβαίω θα αναλάβω εγώ τώρα τη διεύθυνση τη συζητήσεω και έχουμε τώρα τι ερωτήσει. Ο κύριο Σαΐν πρώτο. Ευχαριστώ. Έχω να πω το κυρία Φλότρ. Ανεξαρτήτως προελεύσεως των παθόντων πρέπει να μιλούμε για τέτοιες ανθρωπιστικές τραγωδίες και ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βεβαίως τη δική της γνωστή ιστορία και σε ολόκληρο τον κόσμο σημειώνονται τραγωδίες που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν αν είχαμε διδαχθεί από το παρελθόν. Τα θύματα είναι συχνά μητέρες και παιδιά. και η φωνή τους πρέπει να ακουστεί εδώ. Θα σας παρακαλέσω να μεταβείτε επιτόπου, να δείτε με τα μάτια σας την κατάσταση αυτή. Εγώ είμαι βουλευτής του Gaziantep, όπου, στο νότο της Τουρκίας, όπου υπάρχουν τρεις καταβλισμοί προσφύγων. Είδαμε μάλιστα πριν ορισμένες φωτογραφίες από τους καταβλισμούς αυτούς. Οι Σύριοι αδελφοί και αδελφές μας εκεί έχουν την ε, πρόσθετη ας πούμε ευκολία ότι πολλοί άνθρωποι εκεί από τους δικούς μας μιλούν αραβικά. Όταν αν θέλει κάποιος να μιλήσει μαζί μου μπορεί να έρθει σε επαφή διότι σας άφησα τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου μου εάν ενδιαφέρεστε. Οι διεθνείς σχέσεις στα πλαίσια των οποίων συζητείται και αυτό το ενδεχόμενο δημιουργία μιας ζώνης προστασίας, μιας buffer zone. Βεβαίως, όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή σημειώνονται δράματα. Στις 21 Ιανουαρίου, 3 ώρα το πρωί, χτύπησε το τηλέφωνό μου και εγώ βρισκόμουν εκείνη την ώρα στην Άγκυρα με πήραν τηλέφωνο από κρατικό νοσοκομείο στην περιοχή μου και μου είπαν ότι μόλις είχαν φτάσει πολλά παιδιά από τη Συρία, 7 αδελφάκια. που μόλις είχαν χάσει τους γονείς τους σε βομβαρδισμό. Μόνο τα παιδιά επέζησαν, ήταν όμως τραυματισμένα και έπρεπε να εγχειριστούν τάχιστα. Δεν ήταν προετοιμασμένο το νοσοκομείο και δεν είχε τη δυνατότητα Γι' αυτό τα έστειλαν γρήγορα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Γκάζιαντεπ. Όλα τα νοσοκομεία ήταν υπερπλήρη. Έφτασε η ώρα αυτά το πρωί για να μπορέσουμε να ξεσηκώσουμε τους χειρουργούς από τα κρεβάτια τους και να τους στείλουμε στα νοσοκομεία. Τελευταία στιγμή σώθηκαν ορισμένα από τα παιδιά αυτά, χάρη στη χειρουργική επέμβαση. Αυτά είναι δράματα τα οποία ζουν πολλά παιδιά από τη Συρία. Χάρη στο τηλεφώνημα αυτό στις 3 ώρα το πρωί όπως εξήγησα, σώθηκε το, σώθηκαν τα παιδιά αυτά. Μετά βρήκαμε κάποιους συγκινήσεις τη γιαγιά και ένα θείο. Και έτσι παραδώσαμε τα παιδιά σε αυτούς. Άλλο πάλι ήμουν στην Άγκυρα, ξαναχτυπάει το τηλέφωνο με 9 η ώρα. Με παίρνουν τηλέφωνο κάποιοι σύροι. ακούω ε, στο βάθος φωνές. Ένα κοριτσάκι 7 χρόνων είχε μπορέσει και πέρασε τα σύνορα βαδίζοντας δύο μέρες, αλλά δεν μπορούσε, α, δεν μπορούσε να συνενοηθεί στον καταβλισμό. Ήταν νέες κοπέλες και κάποια νέα κοπέλα ήταν μάλιστα έγκυος. Λάβαμε μέτρα, βρήκαμε θέση για τα παιδιά αυτά. Ήδη είχαν αρχίσει οι οδύνες του τοκετού του κοριτσιού αυτού. Τη στείλαμε με νοσοκομείο, ε, συγγνώμη, με αυτοκίνητο στο κρατικό νοσοκομείο του Νιζίπ αλλά δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη η πέμπτη της εγκυμοσύνη. Και έπρεπε να γίνει αμέσως και σαρική τομή. Μιλώ τώρα ε, για την μητέρα των παιδιών αυτών. Όμως το νοσοκομείο δυστυχώς δεν διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Τέλος πάντων το παιδί γεννήθηκε ευτυχώς. Αλλά δυστυχώς τελικώς δεν επέζησε. Λόγω της ταλαιπωρίας, της πορείας εκείνης. Σας τα λέω αυτά γιατί θέλω εν τέλει να καταλήξω το εξή. Τα πράγματα αυτά, τα δράματα αυτά παίζονται όταν οι φίλοι μας στην Ευρώπη βρίσκονται στα αναπαυτικά τους και ζεστά τους κρεβάτια. Γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Οι συνάδελφοί μας από την Ευρωβουλή χθες φάνηκαν πολύ αναστατωμένοι για τα όσα γίνονται στο πάρκο Γκεζί Σήμερα μιλούμε για ένα πραγματικό ανθρωπιστικό δράμα και στρέφομαι γύρω μου και βλέπω μοναχά δύο ευρωβουλευτέ. Τον κύριο Βαλένσα και την κυρία Παπαδοπούλου, η οποία όμως βλέπω ότι έφυγε πάλι. Και αυτό ήταν. Εγώ θέλω να σημειωθεί αυτό στο πρακτικό σήμερα και το πρακτικό αυτό να σταλεί το συντομότερο δυνατό στους συναδέλφους ευρωβουλευτές ώστε τουλάχιστον ε, να διαβάσουν τα όσα συμβαίνουν στην Συρία. Ευχαριστώ κύριε Σαΐν. Ε, το βίντεο σας διαβεβαίω έχει καταγράψει τις παρουσιάσεις και, ε, του κύριου Χατύπ και θα τη διαδώσουμε και θα τη διαβάσουμε σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε είναι μέλη της Μικτής Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής είτε δεν είναι αυτή. Έχω να κάνω ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, για την υποδοχή σύρων προσφύγων στην Ευρώπη. Το έχουμε ξανασυζητήσει από την αρχή της σύγκρουσης αυτό επανελειμμένα. Γνωρίζουμε ότι οι Σύροι πρόσφυγες ε, τυχάνουν πολύ διαφοροποιημένης υποδοχής. Στη Σουηδία περίπου καλά τους δέχονται, στη Γερμανία λίγο καλύτερα και αρκετά χειρότερα στις υπόλοιπες χώρες και είναι και δύσκολο να διαβούν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης οι Σύριοι πρόσφυγες. Περίπου καταφέραμε στο τελευταίο ψήφισμα μας να εντάξουμε την ιδέα ε, χορήγησης ε, προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής ε, εισρωής. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί κάλλιστα να προσαρμοστεί στην κατάσταση. Για λίγες ψήφους χάσαμε. Αλλά το θέμα τίθεται, είναι συγκεκριμένη η πράξη πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια ή την ενδεχόμενη στρατιωτική και άλλη και οικονομική βοήθεια. Είναι ένας τρόπος να αποδείξουμε στην πράξη την αλληλεγγύη μας με το Συριακό λαό σήμερα. Ο κύριος Τεκελίογλου. Teşekkür ederim. Sayın Başkanlar, ε. Σας ευχαριστώ. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, η κατάσταση στη Συρία είναι γνωστή. Ο κύριος Αλχατίμπ την εξήγησε ε, εκτεταμένα, δεν χρειάζεται να επανέλθω στις λεπτομέρειες. Και εγώ ίδιος επισκέφθηκα έναν από τους καταβλισμούς και πραγματικά δεν μπορούμε να, να μείνουμε συγκίνητοι. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον κύριο Αλχατίμπ το εξή. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σχέδιο ειρήνης, δεν μπορεί να μείνει ε, ασυγκίνητη μπροστά στα όσα συμβαίνουν. Οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίε. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε παρόμοιες περιπτώσεις ε, άργησε να ενεργήσει και ε, έχει αποκτήσει έως και ένα σύνδρομο. Ε, έχουμε καθυστερήσει εμείς απέναντι στη Συρία, ναι, εν μέρη, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και ελπίζω πως η διάσκεψη της Γενέβης θα οδηγήσει σε κάτι θετικό. Όμως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρες που είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, των Ηνωμένων Εθνών. Πολλοί θα ήθελαν να επηρεάσουν, να μπορέσουν να επηρεάσουν την Κίνα και τη Ρωσία, αλλά και το Ιράν. Δεν άκουσα να έκανε κάτι ε, ε, ιδιαίτερο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως εμένα να μου διέφυγε, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Η Νότια Αφρική, για παράδειγμα, ε, υπήρξαν, ε, επιβλήθηκαν πολύ σοβαρές κυρώσεις ε, στο νοτιοαφρικανικό καθεστώς που υποχρεώθηκε να συνομιλήσει με τον Νέλσον Μαντέλα. Όμως τέτοιου είδους κυρώσεις δεν έχουν εφαρμοστεί για τη Συρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο ενός, μιας πολιτικής λύσης. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση και στη Βοσνία η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε παρέμβει με κάποια καθυστέρηση. Αφού είχαμε ζήσει πολλές τραγωδίες, ελπίζω πως ε, και ε, το πρόβλημα της Συρίας ε, θα λυθεί χωρίς απεραιτέρω καθυστέρηση. Ένα άλλο ερώτημα τώρα που έχω προς τον κύριο Αλχατίμπ. Ο κατακαιρματισμός της Συριακής Αντιπολίτευσης μας ανησυχεί. Εάν μπορείτε να με καθησυχάσετε θα ήταν πολύ ωραία, αλλά ακούγονται πολλές φωνές από την Συριακή Αντιπολίτευση. Οι οργέτες ε, το, της αντιπολίτευσης κατά κάποιο τρόπο ε, είναι πολύ και διάφοροι και αυτό ε, δημιουργεί πρόβλημα στην, στον αγώνα κατά του τύραννου Αλάσαντ. Να πω κάτι ακόμα για τη Συρία. Το πρόβλημα μια θρησκευτική σύγκρουση είναι το λιγότερο, το μικρότερο κακό ε, αυτή τη στιγμή πρέπει να αγωνιστούμε για πολιτική ελευθερία. Οι Σύριοι φίλοι θα πρέπει να αφήσουν κατά μέρο τον φόβο σε σχέση με τις θρησκευτικές τις συγκρούσεις και να προχωρήσουν προς δημοκρατική και πιο ελεύθερη λύση για τη Συρία. Ευχαριστώ. Κύριε Μετόζοκλου, θα νομίζω πως είναι καλό να θυμίσετε ποιες είναι οι κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συριακό καθεστώς, γιατί η Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις, έχει πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας, ε, όπως καταλαβαίνετε παρεμποδίζεται στις πολιτικές της πρωτοβουλίες λόγω ε, της έλλειψης ομοφωνίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου, ακόμα και αν διαπιστώνω πως ε, οι πιο πρόθυμες χώρες για να παρέμβουν και με στρατιωτικό τρόπο, όπως η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, έχουν επιτρέψει την αναγνώριση του συνασπισμού σε προσώπου του Συριακού λαού, που, πράγμα που είναι σημαντικό. Και είπαμε να άρουμε και απο πρώτη 1η σε 8 το εμπάρκο στα όπλα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν πολλές χώρες. Εγώ είμαι Γαλλίδα και Καταλαβαίνω την πολιτική της χώρας μου και των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, αλλά η Γαλλία είναι πάρα πολύ δραστήρια. Έχει αναπτύξει διόδους στήριξη της αντιπολίτευσης στη Συρία. Και μάλιστα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Αλχατίμπ, Η εποχή μετά Ασάντ προετοιμάζεται από τώρα. Υπάρχουν απελευθερωμένες ζώνες όπου όμως υπάρχει μέγα διακύβευμα αρχίσει να οικοδομείται η μελλοντική διοίκηση του κράτους μετά τον Ασάντ, γιατί πιστεύω πως αυτό ραβάζοντας όλους τους φορείς σε αυτή την προοπτική μετά Ασάντ θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη δυναμική που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε το δράμα μέσα στο οποίο είμαστε βυθισμένοι σήμερα με την έλλειψη προοπτικής δηλαδή και την ε, και τους, τις ουρές προσφύγων και δράματος που εκτείνεται στο άπειρο, εκτείνονται στο άπειρο. Άρα λοιπόν σήμερα βλέπετε με τη βοήθεια τη διεθνή, με τη βοήθεια της Ευρώπης πώς θα μπορέσει να, να οικοδομηθεί μια πρώτη δίκηση μετά τον Ασάντ ώστε να μπορέσει να επανεγκαθιδρυθεί μια ζωή με κάποια κρατικά έμβρια για να προετοιμαστεί η συνέχεια. Η κυρία Ντανίσογλου. Α, έφυγε από την αίθουσα. Ο κύριος Ραμαζάνογλου. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε σχέση με τα όσα είπατε, εγώ θέλω να κάνω την εξής απλή διαπίστωση και μετά έχω δύο ερωτήσεις στον κύριο Ελχατίμπ. Η, ε, η, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία βασίζεται πολύ στην ρωσική θέση. Ε, ο, ο Αλασάντ χρησιμοποιεί χημικά όπλα και αυτά εξ αρχή. Ωστόσο αυτό δεν μετέβαλε τη θέση των Ρώσων. Η διεθνή κοινή γνώμη λέει ότι πρέπει να φύγει ο Ασάντ και έχουμε την εντύπωση ότι περιμένουμε διαρκώ την έγκριση της Ρωσίας. Από τη μια πλευρά λέει λοιπόν η Ρωσία ότι δεν είμαι κατά της αποχώρησης του Ασάντ, αλλά από την άλλη Από την άλλη, την άλλη εμποδίζει την αποχώρησή του. Στη διεθνή κοινή γνώμη λοιπόν προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιο σύστημα θα φτιαχτεί από τη στιγμή που θα έχει φύγει ο Ασάντ. Και η διεθνής κοινή γνώμη δεν θέλει να δει καταφτάνει στη Συρία ε, στην εξουσία άνθρωποι, οι οποίοι θα επηρεάζονται από την Αλκάιντα. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αλχατίμπ. Στην κοινή γνώμη γίνεται λόγος από καιρού καιρών ε, γίνεται λόγος για την επιρροή της Αλκάιντα. Ποια είναι η κατάσταση της Αλκάιντα στην Συρία. Είναι σημαντική, έχει επιρροή όντως. Άλλη μια ερώτηση. Οι δυνάμεις του Ασάντ έχουν συνεργαστεί με την Χεσμολά για να καλυφθεί το κενό που ήταν στα χέρια της αντιπολίτευσης και για να πάρουν την πόλη Συγγνώμη, για να, για να ξανακατακτήσουν τις πόλεις που ήταν στα χέρια της αντιπολίτευσης και αρχίζουμε να σκεφτούμε σκεφτόμαστε πως ο Ασάντ μάλλον είχε φύγει από την... Ε, είχε εγκαταλείψει την εξουσία βράχη πρόθεσμα, μήπως... Ε, ήθελε λοιπόν να διατηρήσει ένα κομμάτι της επικράτειας όπου θα μπορούσε να καταφύγει και να προχωρήσει προς έναν κατακαιρματισμό της Συρίας σκοπεύει να δημιουργήσει ένα κομμάτι, μια περιφέρεια που θα μπορεί να είναι αυτόνομος. Αυτά. Σας ευχαριστώ από τώρα κύριε Αλχατίμπη για τις απαντήσεις. Ο κύριος Γκύρου. Ah, euh. Μάλλον να θέσω και εγώ την ερώτησή μου πριν να παρέμβεστε. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ακριβώ επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την Ευρωμικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή, την παρουσία ενό εσύριου ηθήνοντο, είναι σημαντικό να συζητήσουμε και για του Κούρδου σε αυτή τη σύγκρουση. Γιατί βέβαια υπάρχει φυσικά σχέση ανάμεσα στην ειρηνευτική διαδικασία που έχει ξεκινήσει στην Τουρκία και τα διακυβεύματα της πολιτικής που ασκούν οι Κούρδοι στη Συρία, ποια είναι η κατάσταση σήμερα, τι μπορούμε να περιμένουμε για αυτές τις ζώνες που είναι αρκετά πολύ άριθμες στα τουρκοσυριακά σύνορα που είναι υπό τον έλεγχο του κουρδικού ε, ε, ε, πληθυσμού. Ξέρω σε ποιον θέτω την ερώτησή μου. Εσείς κύριε Γκούρ. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, περίπου το ίδιο θέμα θα έφυγα κι εγώ. Ο κύριος Αλχατίμπ είπε πολύ, ε, μάλλον περιέγραψε σαφώς ε, το, τις διαστάσεις του δράματος που ζει αυτή τη στιγμή η Συρία. Θα ήθελα να τον ήξερα προηγούμενα, νωρίτερα, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες της κατάστασης αυτής στη Συρία ε, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια πολιτική λύση θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν κάπως περισσότερο τα πράγματα. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ανεπαρκής κυρίως από πλευράς της, Ευρωπαϊκής, της διεθνούς κοινότητας, αλλά η επίλυση του Συριακού μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας φυσικά δεν πρόκειται, δεν είναι αρκή. Ίσως θα έπρεπε να γίνει και μια ανθρωπιστική ε, επέμβαση. Ίσως η Δύση ε, να πρέπει να πιστεί να πιστεί η Ρωσία, η Κίνα για τη σημασία μιας ε, παρέμβασης ανθρωπιστικής. Υπάρχουν ε, αντιφατικά συμφέροντα, αλλά υπάρχει ένα άλλο σημαντικό θέμα, είναι η μετά Ασάντ εποχή. Τι θα γίνει μετά τον Ασάντ... και συμμερίζομαι τα όσα είπε ο κύριος Τεκελιόγλου. Δεν ε, έχουμε να κάνουμε μόνο με τις ε, θρησκευτικές συγκρούσεις. Ε, υπάρχουν τα προβλήματα των μειονοτήτων. Υπάρχουν το, δηλαδή Αρμένοι, Κούρδοι που είναι συγκεντρωμένοι σε συγκεκριμένες περιοχές και ζουν σε μεγάλες πόλεις όπως η Δαμασκόζη, το Χαλέπι, ένα σωρό ερωτηματικά δηλαδή. Και η ε, Συριακή Αντιπολίτευση θα θέλαμε να καταφέρει να δημιουργήσει μια δημοκρατική Συρία αύριο. Αλλά υπάρχουν οι Δρούζοι, οι Κούρδοι, οι Αρμένοι. Οι Αρμένοι θα πρέπει να μπορέσουν όλοι να αντιπροσωπεύονται μέσα στο πλαίσιο αυτής της αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή όμως, μέχρι σήμερα δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Υπάρχει επιρροή διαφόρων ε, φανατικών Ισλαμιστικών ομάδων που θα θέλαν να έχουν περισσότερη εξουσία στο πλαίσιο της αντιπολίτευσης και όλα αυτά αποδυναμώνουν την ε, Συριακή αντιπολίτευση, κυρίως στο επίπεδο της διεθνούς κοινή γνώμης. Όσον αφορά τους Κούρδους, φυσικά είμαστε ευαίσθητοι για το θέμα αυτό, αλλά έχουμε και μια ευαισθησία σε σχέση με όλους τους λαούς που ζουν στη Σύρια. Δεν έχουμε μόνο προσέγγιση για τους Κούρδους. Ναι. Ε, η Συρία είναι ένα σύνολο και ολόκληρος ο Συριακός λαός, όποια και αν είναι η, προέλευσή του, Κούρδοι, Δρούζοι, Αρμένοι, ε, Ασσύριοι και ένα σωρό άλλοι, ε, πρέπει να μπορούν ε, από μόνοι τους να καθορίσουν το μέλλον τους. Πολύ λίγα έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Έχουν φτιαχτεί όντως καταβλισμοί από την Τουρκία, αλλά Υπάρχει και μια άλλη κατάσταση στις περιφέρειες όπου ζουν οι Κούρδοι. Υπάρχει εμπάργο, το οποίο έχει εφαρμόσει το Συριακό καθεστώς και η βοήθεια δεν φτάνει μέχρι εκεί στις κουρδικές περιοχές. Γνωρίζουμε ότι ο πληθυσμός εκεί αυξάνεται σαφώς το τελευταίο καιρό. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός κατά 200-300%. Οι Κούρδοι βοηθούν αυτούς τους εκτοπισμένους και την περασμένη εβδομάδα μια αντιπροσωπεία ε, τους ήρθε στην Άγκυρα, είχε επαφές με διάφορα υπουργεία και εκπροσώπους ε, της περιοχής, της περιφέρειας μάλλον, ε, Γκάζι Αντέμπ. Και θα ήθελαν ο ελεύθερος συριακός στρατός να άρει το εμπάργο που ισχύει μέχρι στιγμής σε αυτές τις περιοχές για να μπορέσει να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Έγινε μια πολύ, είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Ε, ήθελαν ε, να φτιάξουν δύο καταβλισμούς. Έχουν δύο προγράμματα για καταβλισμούς. Ένα στην περιφόρεια του Ζιζρέ για να μπορέσουν να υποδεχθούν τους ε, Σύριους που έχουν εκτοπιστεί χωρίς καμία διάκριση, έτσι ώστε όλοι οι Σύριοι να μπορέσουν ε, να ε, εγκατασταθούν εκεί ειρηνικά και με ασφάλεια. Έχουν ε, τη στήριξη της, μάλλον χρειάζονται τη στήριξη της Τουρκίας, της Συριακής Αντιπολίτευσης αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Οι Σύριοι Κούρδοι αγωνίζονται για μια δημοκρατική Συρία. και νομίζω πως ε, τίνουν να ενεργήσουν με την Συριακή Αντιπολίτευση, αλλά θα πρέπει για το λόγο αυτό η Συριακή Αντιπολίτευση ήδη να λάβει υπόψη της το σύνολο των λαών που ζουν στη Συρία και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην υπάρξει θρησκευτική σύγκρουση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα δικαιώματα της χριστιανικής κοινότητας στη Συρία, πράγμα που θα διεύρυνει και όλα στη βάση της αντιπολίτευσης. Και αυτή, ε, αυτός ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης, όπως είπε και η Ελέν, θα ήταν αποτελεσματικό για να φανεί στις απελευθερωμένε περιοχέ τη Συρίας ότι υπάρχει μια νέα προσέγγιση και μια νέα προσπάθεια. Ξέρω πω μακρηγορώ, αλλά ήθελα να προσθέσω ακόμα ένα σημείο πως ε, δηλαδή υπάρχει μια ανθρωπιστική βοήθεια που συνεχίζεται στη Συρία, αλλά θα πρέπει ε, κυρίως να υπάρξει μια παρέμβαση στρατιωτική. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δεμερκυρά. Ο κύριος Οκτάη σας ε, περιέγραψε τα όσα γίνονται στη ε, Τουρκία. Στο νομό Μαρντίν, ε, δίπλα σε ένα μοναστήρι, δημιουργήθηκε ένας καταβλισμός με χωρητικότητα 3.000 και είχε στόχο να υποδεχτεί τους Ασυρίους, Ασυροχαρδαίους. Ε, κοντά σε, μια μονή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα αιτήματα. Φαντός αυτός ο καταβλισμός μπορεί απολύτως να τους υποδεχθεί ε, ε, δίπλα στο μοναστήρι τους. Υπάρχουν ε, δυνατότητες. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν απευθύνεται σε μία κοινότητα, είπαμε, ούτε σε μία θρησκεία. Ε, ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα όλων. Το λόγο έχει ο κύριος Ιουσίκ. Ευχαριστώ κύριε Συμπρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, υποβάλλω τα σέβη μου. Εγώ θυμάμαι τη σφαγή στη Χάμα, τότε ήμουνα στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Ο Ασάντ Πατήρ είχε στείλει τα τάγκς, ε, περικύκλωσε την πόλη και ε, κατακρεούργησε τον τόπο. Εγώ τότε ήμουν μαθητής, θα θυμάμαι αυτά, ε, ήμουν στο γυμνάσιο. Η Ευρώπη εισηγεί ηχθείως και στον παγκόσμιο τύπο επίσης πουθενά δεν το είδαμε. Ε, ο τύπος στην Τουρκία επίσης ήταν υποποίηση ένα μονόστιλο, κάπου ένα μικρό άρθρο είδα σε ένα ισλαμιστικό περιοδικό. Εγώ ε, στο αρχείο μου έχω ακόμα τις φωτογραφίες από εκεί και θυμήθηκα τη σφαγή της Χάμα ε, με όσα γίνονται σήμερα. Οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, κρίμα που δεν είναι σήμερα εδώ, θα έπρεπε. Εχθές έγινε λόγος ε, για τις διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίμ ενώ στη Συρία οι νεκροί ξεπερνούν τις 100.000 και συνεχίζεται η βιαιότητα και οι αγριότητες και η ε, απουσία των ευρωβουλευτών. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά που τα εφαρμόζουμε και στην περίπτωση της Συρίας. Ε, εδώ βλέπουμε τα προβλήματα και τις ελλείψεις. Ακούγεται από όλους ε, κριτική. Η κυρία Φλότρ μίλησε για το κουρδικό ζήτημα αλλά και στο εσωτερικό του κόμματος ΑΚΕΠΕ υπάρχουν κουρδικής καταγωγή βουλευτές. Δεν είναι ε, οι βουλευτές μόνο του ΜΠΕΝΤΕΠΕ Κούρδοι που έχουν κουρδικές ευαισθησίε και στο δικό μας κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Ισικ, λέει ο συμπρόεδρος. Νομίζω ότι ναι, έχουμε τρει-τέσσερι Κούρδου αυτή τη στιγμή παρόντε, δεν υπάρχει καμία διάκριση ανεξαρτήτω κομμάτων. Ναι, η κυρία Φλότρ μπορεί να είχε να κάνει μια ερώτηση στον κύριο Αλχατίμπ, δεν ξέρω, για τη Συρία. Και εγώ βουλευτή στο ΑΚΠ είμαι και έχουμε και πολλού κουρδική καταγωγή βουλευτέ, κυρία Φλότρου, και στο δικό μα κόμμα. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Σογιάν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συμπρόεδροι, σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια στην Τουρκία, ε, βεβαίως γίνονται πολλές προσπάθειες, πολύ μεγάλη οργάνωση πολύ καλή οργάνωση ε, και η Τουρκία πραγματικά ανταποκρίνεται στις περιστάσεις. Σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, η Τουρκία μπορεί να δώσει μαθήματα ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τετραπλάσιο κατακεφαλήν εισόδημα σε σχέση με την Τουρκία και παρόλα αυτά η Τουρκία απέδειξε ε, μία άψογη αλληλεγγύη. Και έχει να διδαχθεί, πιστεύω, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη από αυτή την προσπάθεια της Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανθρωπιστική βοήθεια, η Ευρώπη αντί να δώσει ανθρωπιστική βοήθεια αποφάσισε να στείλει όπλα στη Συρία. Αυτό με εξέπληξε πρέπει να σας πω πάρα πολύ. Στη Συρία υπάρχει μια ηγεμονική ε, δύναμη, μια εξουσία που ενισχύθηκε ακόμα πιο πολύ από τη στάση της δύση. Και σήμερα το καθεστώς έχει έρθει σε αμυντική θέση. Υπάρχουν και σαλαφιστές μαχητές εκεί που ε, αγωνίζονται κατά του καθεστώτος. Υπήρχε η Αλκάιντα, η Αλούσρα και διάφορα άλλα παρακλάδια και ε, σφαγή γίνεται εκεί και τους αλεβίτες και τους χριστιανούς αυτοί τους φάζουν. Τους έχουν περικυκλώσει από έναν ε, ε, κυρίαρχο σουνιτισμό. Και η Ευρώπη πιστεύω εθελοτυφλή. Δεν θέλει να δει αυτό το κίνδυνο. Οι χώρες όπως η Τουρκία, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία κτλ. Είναι επίσης χώρες διέλευσης για την βοήθεια, τα όπλα δηλαδή που στέλνονται εκεί. Και θέλω να ρωτήσω, είναι άραγε δημοκρατικές χώρες το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία και δεν το έχουμε πάρει είδηση. Διερωτώ με. Και θέλουμε μετά να υποστηρίξουμε ένα Ισλαμιστικό καθεστώς που θα εγκαθιδρυθεί αν ρίξουν τον Άσαντ. Αυτό θέλουμε. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω την κατάσταση σήμερα. Ε, ε, ε θέλω να πω το εξής τώρα. Ο κύριος Χατίπ μίλησε για ένα τρομοκράτη, κράτος τρομοκράτη που εδώ και 50 χρόνια τους καταπιέζει. Πριν από τρία χρόνια η κυβέρνηση Ερντογάν συνεδρίαζε και συνομιλούσε με το καθεστώς αυτό. Έκτοτε τι έγινε, δηλαδή τι άλλαξε, τι ανετράπη. Και εγώ προβληματίζομαι. Υπήρξαν αραβικές δημοκρατίες εκεί γύρω στην περιοχή και δεν το είχαμε αντιληφθεί 50 χρόνια τώρα. Η Συρία είναι ένα καθεστώς καταπιστικό βεβαίως, κατασταλτικό, αλλά ήταν μια χώρα σχετικά κοσμική, μη θεοκρατική. Τώρα το Ιράκ έχει κοπεί στα τρία. Κινδυνεύει και η Συρία ε, και ε, κινδυνεύει να γενικευθεί η σφαγή στη Συρία και τέλος και στα Πέριξ και θα πρέπει, λέμε, να βρούμε μια λύση μέσα σε ένα διάλογο. Συμφωνώ. Αλλά η λύση βρίσκεται στη Γενέβη. Ναι, βεβαίω να ε, συγκληθεί η δεύτερη διάσκεψη τη Γενέβη, λεγόμενη Γενέβη 2. Δεν θα πρέπει να υποδαβλίζουμε αυτό τον εμφύλιο πόλεμο, δεν βοηθάει κανένα, δεν εξυπηρετεί κανένα και ενέχει και τον κίνδυνο περιφερειακή σύραξη γενικότερη. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί μια πολιτική λύση και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη αλλά και άποψη του κόμματός μας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ο καθηγητής ο Γιάν μίλησε, σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Ε, δεν θέλει κανείς άλλος το λόγο. Όπως βλέπω είναι πάρα πολύ λίγοι οι Ευρωπαίοι βουλευτές που παρευρίσκονται σήμερα. Πολύ κρίμα και πολύ περίεργο το βρίσκω, λέει ο κύριος Ντεμίρ Κιράν, συμπρόεδρος. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αν το χρόνο σε ευρύτερη ομίγυρη, γιατί σήμερα συζητούμε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ τραγικό. Ο κόσμος χάνεται ε, και αδιαφορούν πλήρως οι πάντες. Αυτό πραγματικά μας ε, θλίβει και μας λυπεί βαθύτατα. Και είμαι βέβαιος, κυρία Πρόεδρε, ότι συμμερίζεστε αυτές τις απόψεις μας. Αυτά. Να δώσω το λόγο στην κυρία Φλότρο για την παρουσία των Ευρωβουλευτών και τον αντίκτυπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της συνεδρίασης αυτής, ε, σας είπα ότι υπερβαίνει τη συγκεκριμένη, τα συγκεκριμένα πλαίσια της σημερινής μας συνεδρίασης. Γιατί έχουμε και συνέντευξη τύπου μετά το πέρας της συνεδριάσεως, στην οποία θα επιθυμούσα να μπορέσει να συμμετάσχει και ο κύριος Αλχατίμπ γιατί το δικό του λόγο θέλουμε να ακούσουμε σήμερα η δική του φωνή είναι σημαντικό να ακουστεί σήμερα στην Ευρώπη ε, τα εδώ διαμευθέντα έχουν ε, μαγνητοσκοπηθεί και θα διαβιβαστούν. Ξέρετε ότι μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει στις συνεδριάσεις και με άλλους τρόπους πέρα από τη φυσική και άμεση παρουσία στην αίθουσα που είναι το βασικό θα έχει αντίκτυπο και θα υπερβεί το σημερινό πλαίσιο η συνεδρίασή μας. Να είστε βέβαιοι, μην αμφιβάλλετε γι' αυτό. Ο κύριος Γιάν, και πριν δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, θέλω να πω στον κύριο Γιάν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία. Ο πρώτος, ο παριθμόν ένα. Τι χαμογελάτε, τι μηδιάτε. Αυτό δεν λέμε από προηγουμένως. Για τη χρηματοδότηση είπαμε δεν είναι επαρκές, το ξέρουμε. Χρειάζεται ε, μια σοβαρή και αποτελεσματική πολιτική προοπτική και πρωτοβουλία. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως περιορίζεται ε, και έχει ένα εμπόδιο που είναι η ομοφωνία στο Συμβούλιο. Θέλω να το επαναλάβω. Είναι γεγονός. Βέβαια αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από την υπόθεση ότι είναι υπαριθμόν ένα δωρητής η Ευρώπη της ανθρωπιστικής βοήθειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Τώρα, εγώ ίδια είμαι εκείνη που λέγω ότι ε, η ανθρωπιστική βοήθεια δεν αρκεί. Θα πρέπει να περάσει ε, και σε δυνατότητα υποδοχής προσφύγων, όχι μόνο χρήματα ή πολιτικές πρωτοβουλίες. Όλα αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα πιστεύω και η ενίσχυση των δυνατοτήτων διεθνούς προστασίας και υπεράσπισης και της αντιπολίτευσης Συρία σήμερα συμπεριλαμβανομένη στις προμήθειες όπλων και ελεγχόμενων. Ξέρουμε γιατί θα περάσει μέσα από τον ελεύθερο Συριακό στρατό και τον στρατηγό τον κύριο Ιντρίς αν δεν απατώμε. Και ε, έχουμε τα εχέγγυα, ε, θα πρέπει να έχουν να μην φτάσουν τα όπλα αυτά ε, στα χέρια εκείνων που δεν θέλουμε να φτάσουν. Ε, αλλά να μην έχουμε και μια αδράνεια και μια απάθεια ε, της διεθνούς κοινότητας. Είναι γνωστά όλα αυτά. Αν μη τι άλλο, ε, θα πρέπει να αναγνωρίζουμε μερικά στοιχεία ανάλυσης κατάστασης, αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει κανείς. Τώρα, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, παρακαλώ. Είναι σημαντικό να ξαναλάβετε το λόγο αυτή τη στιγμή. για να μας πείτε με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από μια θέση που φαίνεται στάση αναμονής ενδεχομένως από πλευράς πολιτικής γιατί περιμένουμε και προσευχόμαστε να γίνει η Γενέβη 2 επιτέλους κάποια στιγμή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ε, να προτείνουμε στα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο για να είμαστε πιο δυναμικοί και πιο δραστήριοι και παρόντες για την πολιτική επίλυση αυτής της σύραξης. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι μου θέτεται μία περίπλοκη και δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη και περίπλοκη διότι αντιμετωπίζουμε μία περίπλοκη κατάσταση. Και ιδίως όταν αντιμετωπίζουμε μάλιστα και την ύπαρξη ενός αριθμού χωρών μελών που είτε μας αρέσει είτε όχι έχουν διαφορετική προσέγγιση. Μιλούμε για διαφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είναι αληθές. Διαφορές υπάρχουν και μέσα στην διεθνή κοινότητα. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής κυρία Πρόεδρε που είναι ότι πιστεύουμε σε πολιτική λύση. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Παρακολουθώ τη συζήτηση και διαπιστώνω ότι όλοι εδώ συμφωνούμε για τη σημασία της πολιτικής λύσεως. Βέβαια, υπάρχουν πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια και δεν μιλώ πάλι για την ενίσχυση που δίνουμε. Είπατε εσείς κυρία Πρόεδρε ότι είμαστε ο πρώτος δωρητής. Τι διαφορά έχει αν έχουμε δώσει 1,2 δις η Τουρκία 1 εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσο, άλλο 1 δισεκατομμύριο, δεν ξέρω. Αλλά τι νόημα έχει. Πρώτα πρώτα αυτό που θέλουμε είναι να συμφωνήσουν οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι για μια λύση. Και μετά να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα μέρη. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πείσουμε να αποκτήσει η αντιπολίτευση μια πιο ενιαία θέση. Βεβαίω μιλούμε και για το καθεστώς. Αλλά υπάρχει ένα θέμα και με την αντιπολίτευση. Υπάρχουν πρωτοβουλίες, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ εδώ, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε για να εμπλέξουμε έστω και έμεσα και άλλους φορείς, άλλους actors. Συνεργαζόμαστε στενά με την Αίγυπτο σε μια προσπάθεια να δραστηριοποιήσουμε την πρωτοβουλία Μορσή, το όνομα του Αιγυπτίου Πρόεδρου. Είπατε κυρία Πρόεδρε ότι οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι στραμμένες προς τα εμπρός. Ναι, η η επόμενη μέρα είναι πολύ σημαντική. Αλλά αυτή θα καθοριστεί από το τι κάνουμε σήμερα και από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ένα πράγμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι αυτό που έδειξε η κρίση αυτή δεν είναι μόνο το θάρρος του Συριακού λαού, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι αυτοί δεν φοβούνται πλέον, είναι και η ελεγγύη που είδαμε εντός της Συρίας μεταξύ των Σύρων Ελπίζω ότι ο Μωάς θα συμφωνήσει. Το ίδιο η κρίση αυτή ε, έδειξε και έναν ε, αριθμό τοπικών θεσμών που έχουν αναπτυχθεί και ιδίως στο Βορρά προσπαθούμε εμείς να ενισχύσουμε αυτές τις τοπικές δομές, τα τοπικά συμβούλια, διότι πιστεύουμε ότι στο μέλλον αυτά θα κληθούν να παίξουν μείζωνα ρόλο στην μελλοντική Συρία και ένας αριθμός πρωτοβουλίων, πρωτοβουλίων συγγνώμη, μέσω της Τουρκίας είναι σημαντικός για να ενισχυθούν αυτά τα τοπικά συμβούλια. Αρκούμε σε αυτά τα σχόλια κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μποτόσοχλου. Το λόγο θα δώσω τώρα στον κύριο Ντεμπράουερ για να επανέλθει στην ανθρωπιστική βοήθεια και επειδή έχουμε την τον επιτετραμένο τις εξωτερικές ε, υποθέσεις κ. Αλή που είναι, ε, όπως είπα, επιτετραμένος για τις εξωτερικές σχέσεις του, του Κουρδικού Συμβουλίου. Τρεις παρατηρήσεις. Η ερώτησή σας πριν από λίγο, κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά την αλληλεγγύη για την ε, υποδοχή και την ανάληψη ευθύνης για τους ανθρώπους που είναι εκτοπισμένοι και τους πρόσφυγες. Ε, περιλαμβανόταν στο θέμα των δηλώσεων της 27ης ε, ε, Απριλίου θα μπορούσαμε να προβλέψουμε περισσότερο μια προσπάθεια εγκατάστασης και όχι προσωρινής υποδοχής. Ο ύπατος εκπρόσωπος για τους πρόσφυγες κ. Γκουτιέρες του ΟΗΕ στη συμφωνία με την Επίτροπο Μάνστρομ προβλέπουν σύντομα το διοργάνωση μιας διάσκεψης κατά τη διάρκεια της οποίας ε, όχι μόνο τα κράτη-μέλη της Ένωσης που το επιθυμούν, αλλά και τρίτες χώρες θα μπορούσαν να κάνουν μια προσφορά για την ανάληψη εγκαταστάσεων για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες ε, προσφύγων και εκτοπισμένων στις ε, γειτονικές χώρες, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εξή. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης, συμφωνώ αλλά μην ξεχνάτε ότι ε, είναι περιορισμένη η δυνατότητα σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που εκτοπίζονται και που μετακινούνται αυτή τη στιγμή και όσον αφορά όσους βρίσκονται στους καταβλισμούς στο Ζαταρί και στην Τουρκία η πρώτη επιθυμία είναι φυσικά να μπορέσουν να περιστρέψουν στα σπίτια τους όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τώρα, σε σχέση με τα όσα είπε ο συνάδελφος με το Σοχλού για την μέρα μετά, θα πρέπει από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που θυμήσατε πω σε αυτή τη φάση είμαστε οι πρώτοι δωρητέ. Όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι γειτονικέ χώρε πρέπει πραγματικά να μπούμε σε μια προοπτική μια ανθρωπιστική κρίση μακρά. Πολύ μακρά κιόλα. Και μάλιστα ακόμα και αν υποθέσουμε ότι βρεθεί πολιτική λύση, παρατηρούμε αυτή τη στιγμή και νομίζω ο συνάδελφος Οκτάη θα, συμφωνεί, βλέπουμε κάποιες επιστροφές ανθρώπων που είχαν ε, πρόσφυγες δηλαδή, οι οποίοι επανέρχονται στη Συρία, πολύ λίγοι βέβαια, αλλά όταν τους ρωτάμε γιατί ξανάρχονται στη Συρία, συνήθως δυστυχώς είναι γιατί και εκεί φτάνουμε στα όρια της ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι συνθήκες υποδοχής παρά τη στήριξη δεν αρκούν. Δεν είναι ακόμα συνθήκες ασφάλειας. Και λένε τελικά Αφού έτσι κι αλλιώ ε, οδύνει και κίνδυνος, καλύτερα να είναι στη χώρα του τουλάχιστον. Όποια και αν είναι η φιλοξενία που το να του προσφέρθηκε από τις γειτονικέ χώρες. Είμαστε σε μια κατάσταση λοιπόν πολύ μακράς ανθρωπιστικής κρίσης και ότι η ανθρωπιστική βοήθεια της διεθνούς κοινότητας θα πρέπει να εκταθεί σε πολλούς μήνες και χρόνια. Όσον αφορά τη διμερή βοήθεια προς την Τουρκία που ήταν ένα θέμα που έθιξε ο συνάδελφος Ακτάη πριν από λίγο, ένα μεγάλο κομμάτι των ποσών που ανέφερα ε, περνούν από τις οργανώσεις ε, ε, του ΟΗΕ Είτε την είπατε αρμοστή, την UNICEF με την οποία συνεργάζεσαι αυτή τη στιγμή. Μιλήσατε για μικρά ποσά. Ε, ε, συμφωνώ μαζί σας, γι' αυτό και σύντομα θα συγκαλέσουμε συνεδρίαση των κρατών μελών για να δούμε σε ποιο βαθμό συλλογικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη θα μπορέσουν να ενισχύσουν την τεχνική του συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια με τις οργανώσει που είναι παρούσες στην Τουρκία και τις Τουρκικέ αρχές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ, όπως είπα, κατ' εξαίρεση και για λίγα λεπτά, ο εκπρόσωπος του ανώτατου Συμβουλίου των Κούρδων της Συρίας, ο κύριος Ασάν Μοχάμετ Αλή. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να εκφράσω την θέση μας σε σχέση με την κρίση στη Συρία και τις λύσεις που εμείς ε, διαβλέπουμε για την ε, έβρεση διεξόδου. Μιλάμε για καταστροφές στη Συρία και εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι μετά από δύο, δύο χρόνια και τρεις μήνες έχουμε φτάσει στις 100.000 νεκρούς άλλες 100.000 τραυματίες, πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και 5 εκατομμύρια εκτοπισμένοι. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι τα αποτελέσματα ενός πολέμου που διαρκεί εδώ και δύο χρόνια και τρεις μήνες. Εάν συνεχιστεί αυτή η, αυτός ο πόλεμος θα είναι η καταστροφή απόλυτη, μια απόλυτη ανθρώπινη τραγωδία. Γι' αυτό και εξ αρχής επιμείναμε στην εξέβρεση πολιτικής λύσης. Αλλά το βασικό θέμα είναι πώς θα διαχειριστούμε τη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Ασάντ. Εμείς Πιστεύουμε πως η λύση συνίσταται στην ανάπτυξη ενός συριακού έθνους δημοκρατικού με τη συμμετοχή όλων των εθνοτικών ομάδων. Αν δεν καταφέρουμε να αναπτύξουμε μια Συρία δημοκρατική, εάν η νέα Συρία φέρει τη σφραγίδα μιας εθνοτικής ή θρησκευτικής ομάδας, θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες. Η λύση πρέπει να είναι η λύση για όλους τους Σύριους, ώστε όλοι οι Σύριοι να μπορέσουν να εκφράσονται στη νέα Συρία και για να μιλήσω για την κατάσταση των Κούρδων. Υπάρχει μια κατάσταση αρκετά σοβαρή. Στο πλαίσιο όλων των λύσεων που έχουν προβληθεί δεν λαμβάνεται αρκετά υπόψη η σημασία των μειονοτήτων στη Συρία. Η σημασία ε, ε, μειονοτήτων όπως οι Κούρδοι. Είναι απαραίτητο να μην αρκεστούμε στο να θίξουμε απλά και μόνο μια αλλαγή τη εξουσίας, αλλά αλλαγή της φύσης του καθεστώτος και των θεσμών. Διαφορετικά η τραγωδία θα συνεχιστεί. Από ανθρωπιστικής άποψης η κουρδική περιφέρεια που υποδέχεται πάνω από ένα εκατομμύριο Συρίους από την έναρξη της σύγκρουσης, αυτή η ζώνη, αυτή η κουρδική περιφέρεια δεν έχει λάβει ε, ε, καμία ανθρωπιστική βοήθεια από πλευρά των χωρών που υποτίθεται ότι στηρίζουν την ε, Συρία. Από την άλλη πλευρά, αυτές οι περιφέρειες που ήταν περιφέρειες ασφαλή, τις οποίες διαχειρίζονταν οι ίδιοι του, οι Κούρδοι, είναι περιφέρειες οι οποίες έχεραν μια αυτονομία, αυτές οι περιφέρειες μπορούν να αποτελέσουν ένα πρότυπο διαχείρισης ήμασταν σε θέση να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε αυτές τις περιφέρειές μας και ότι είμαστε σε θέση να τις διαχειριστούμε μόνοι μας. Σας ευχαριστώ και πάλι που μας δώσατε την ευκαιρία για να πάρουμε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Επανερχόμαστε στο βήμα τώρα με τον κύριο Κτάη. Θέλετε να απαντήσετε στις παρεμβάσεις που έγιναν. Ο κύριος ε, θα κλείσει αμέσω μετά και θα κάνει και τι παρατηρήσει του και θα απαντήσει στις ερωτήσεις. Κύριε Σοκτάη. E, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τρία είναι ε, τα θέματα στα οποία θα επιθυμούσα να επανέλθω. Στους καταβλισμούς έχουμε μέχρι σήμερα 330.000 ε, πρόσφυγες που είναι υπό την αιγίδα της ΥΠΑ της Αρμοστίας το ΙΕ για τους πρόσφυγες. Ε, Να δεύτερο που ανέφερε η Πρόεδρος για την ενίσχυση, ε, τη βοήθεια που πηγαίνει είτε στη Συρία είτε στην Τουρκία δεν υπάρχει καμία διάκριση, κανένα κριτήριο γι' αυτό. Ε, παράδειγμα, ε, έχουμε το καταβλισμό ε, που είναι για Ασσυρίους, Ασσυροχαλδαίους δίπλα σε μία μονή ε, και σε τακτά χρονικά διαστήματα επίσης δίνουμε βοήθεια σε αποστράτους ε, στρατιωτικούς ε, που υπηρέτησαν στο στρατό του Άσαντ. Ε, βοηθούμε όλους τους πρόσφυγες και επιτρέπουμε και υποβοηθούμε και τον επαναπατρισμό τους. Θα ήθελα όμως να πω το εξή σε σχέση με την Τουρκία. Εκτός των καταβλισμών υπάρχουν προβλήματα. Όχι μέσα στους καταβλισμούς, αλλά με τους πρόσφυγες που δεν διαβίουν σε καταβλισμούς. Και εκεί θα χρειαζόμασταν κάποια ε, καλύτερη συνεργασία και πιο συστηματική βάσει συγκεκριμένων έργων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και projects για τους σύρους πρόσφυγες που δεν έχουν ενταχθεί σε καταβλισμούς, ε, που ε, είναι εκτός των καταβλισμών στην Τουρκία. Και εκεί μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να χρησιμοποιήσουμε την κοινή εμπειρία. Ένα τελευταίο που θέλω να πω στα τουρκο-συριακά σύνορα, ε, από τη συριακή πλευρά, υπάρχουν 10 καταβλισμοί. Συριακοί δεν είναι, είναι από τη συριακή πλευρά των σύνορων, που υποδέχονται από 80 μέχρι 100.000 ε, πρόσφυγες. Γνωρίζουμε ότι είναι ικτρές οι συνθήκες εκεί διαβίωσης των προσώπων αυτών και ε, αποστέλουμε καθημερινώς βοήθεια. Ε, και τρόφιμα, νερό, αλεύρι κτλ. Καλό είναι να δοθεί και ιδιαίτερη προσοχή από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτού του καταβλισμού στη Συριακή πλευρά. Να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι ακριβώ τα σύνορά μα από την πλευρά τη Συρία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Το λόγο θα λάβει πάλι ο κύριο Κατίμπ Αλ-Κατίμπ πιο σωστά για να εξαγάγει τα πολιτικά συμπεράσματα από τη συζήτηση που έγινε γύρω από τα συγκεκριμένα θέματα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ ιδιαίτερος την Πρόεδρο και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις Πρώτον, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκα στην πολιτική διάσταση, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενέκρινε απόφαση που να συμβαδίζει με τη βαρύτητά της. Λάβαμε και το αναγνωρίζω σημαντικότατη ανθρωπιστική βοήθεια και σε αυτήν συμμετέσχουν όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοσημείωτη λοιπόν ανθρωπιστική βοήθεια, το ίδιο ισχύει και για τις Ενωμένε Πολιτείε. Εγώ διαμαρτυρήθηκα στον πρέσβη της Κίνας και τον βεβαίωσα ότι δεν λάβαμε επαρκή ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Κινέζος πρέσβης μας είπε ότι πρόσφερε ένα εκατομμύριο δολάρια και εγώ επέμεινα ότι δεν είναι δυνατόν, αυτό δεν αρκεί. Θα έπρεπε να λάβουμε ένα δολάριο για κάθε Κινέζο πολίτη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τώρα στις διάφορες παρεμβάσεις σας. Θέλουμε να διατηρήσουμε την πίεση επί όλων των μερών για να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι. ακόμα περισσότερο από το καθεστώς, ακόμα περισσότερο από την αντιπολίτευση, μετράνε οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους κάθε μέρα. Η πρώτη στη αποστολή μου είναι να μπορέσω να σώσω ανθρώπους. Εξακολουθώ να είμαι πρόεδρος του Εθνικού Συνασπισμού και αναμένω τις νέες εκλογές για να εγκαταλείψω τη θέση μου. Ο πρόεδρος μένει στη θέση του μέχρι ότου διεξαχθούν νέες εκλογές. Και αναμένοντας, εμένω στην πρώτη στη αποστολή μου, δηλαδή να διασωθούν ανθρώπινες ζωές. Όσον αφορά την προσωρινή προστασία που μπορεί ε, να εξασφαλιστεί. Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό και επικίνδυνο θέμα. Χάνουμε μια ολόκληρη γενεά η οποία δεν έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Κάποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται στην Τουρκία, στην Ιορδανία και στο Λίβανο, αλλά είναι ανεπαρκείς. Προτείνω στις ευρωπαϊκές χώρες να διευκολύνουν την έκδοση προξενικών θεωρήσεων για τους σπουδαστέ που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ιδίως τις ανώτερες σπουδές. Έχουμε ορισμένα στελέχη, τα οποία αισθάνονται βαθύτατη απογοήτευση, διότι δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Τα στελέχη αυτά διαβιούν στους καταβλισμούς χωρίς καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Εγώ έχω σκεφτεί ένα είδος εντό εισαγωγικών υιοθεσία για τα πρόσωπα αυτά. Και να δοθούν επίσης υποτροφίες στους σπουδαστές. Αν κάθε χώρα αναλάβει δεσμευτεί να υποδεχθεί έναν αριθμό σπουδαστών, αυτό ήδη μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση στην Συρία. Γιατί η στέρηση της πρόσβασης στη γνώση είναι ακόμα χειρότερη και από την καταστροφή. Μιλήσαμε και για τους κατοίκους της πόλης Όμς. Πρόσφατα έγινε ολόκληρη γιορτή διότι κάποιοι τους έδωσαν αυγά, τα οποία δεν είχαν δει εδώ και ένα χρόνο. Και άλλα προϊόντα, όπως το αλεύρι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει μια πολιτική πρωτοβουλία που να ενισχύσει την ανθρωπιστική βοήθεια. Όσον αφορά την διέρεση εντός των κόλπων της αντιπολιτεύσεως, νομίζω ότι υπάρχουν διάφορες αποκλήσεις όντως. Ο συνάδελφός μας εξήγησε ότι ο ηγέτης της κινήσής μας εγκατέλειψε τη θέση του. Μόνον εγώ το έπραξα αυτό, διότι, διότι έχω άλλες απόψεις. Ακόμα και η πρωτοβουλία που παρουσίασα εγώ ε, μέσα στα πλαίσια του συνασπισμού δεν υποστηρίχθηκε. Νομίζω λοιπόν ότι καλύτερα θα παίξω τον ρόλο μου απ' έξω. Οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Αμφιβάλλουν οι μεν για τους δε. Διότι δεν είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε επί 50 χρόνια. Δεν είχαμε ούτε τις πιο στοιχειώδεις προϋποθέσεις για να το πράξουμε αυτό έτυχε να συνομιλήσω με συμπατριώτη μου Σύρο και λίγες μέρες μετά με κάλεσαν στο τμήμα διότι του μίλησα. Επίσης υπάρχει και η παρέμβαση πολλών περιφερειακών φορέων. Κάθε χώρα έχει βέβαια τις δικές της προσεγγίσεις και ασκεί Τελευταίες εξελίξεις μέσα στα πλαίσια της αντιπολιτεύσεως έχουν σχέση με εξωτερικές πιέσεις και όχι με τις δικές μας πεπιθήσεις. Η θέση της διεθνούς κοινότητας ενισχύει τις τάσεις αυτές. Στην τελευταία συγκέντρωσή μας εγώ ρώτησα, συνάντηση μάλλον ρώτησα, ζήτησα μάλλον από τους φορείς διεθνούς κοινότητας επιθυμείτε όντως να βοηθήσετε το Συριακό λαό ή όχι διασκέψει επί διασκέψεων και κάθε φορά μας λένε ότι η διεθνή κοινότητα θέλει να βοηθήσει την Συρία, να σχεδιαστεί η βοήθεια. Στα πλαίσια των διασκέψεων των Υπουργών Εξωτερικών κάθε φορά που τίθεται το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας, εγώ ζητώ να μιλήσουμε για υλικό που θα προσφερθεί στους Σύρους. Οι διασκέψεις και συνδιασκέψεις δεν σημαίνουν παρά απώλεια χρόνου και κάθε φορά που σημειώνεται απώλεια χρόνου χύνεται αίμα στην Συρία. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Όλοι διαρωτώνται σήμερα τι θα γίνει μετά την πτώση του καθεστώτος. Σε όλη την πορεία της ιστορίας κανένας υπεύθυνος καθεστώτος δεν έχει προβεί σε παρόμοιες αγριότητες. Άλλοι ηγέτες έχουν καταστρέψει γειτονικέ χώρες. Κανένας όμως ηγέτης δεν εξολόθρευσε τον ίδιο το λαό. Κάθεται, και καταστρέφει τη χώρα του την ίδια. Κανένας υπεύθυνος ηγέτης δεν στρέφει τα βλήματα σκούντ κατά του ίδιου του λαού του. Κανένα ηγέτης δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία που να σκοτώνει παιδιά. Τίποτα δεν υπάρχει χειρότερο από αυτά, από τι αγριότητες που προβαίνει ο Μπασάρα Λάσαντ. Είτε πρόκειται για καθεστώς λαϊκό ή θρησκευτικό, κανένα από τα καθεστώτα που γνωρίζουμε δεν είναι χειρότερο από αυτό που βλέπουμε εκεί. Ο Συριακός λαός έχει ιστορία. Είμαστε η κοιτίδα της ανθρωπότητας. Η γειτονιά όπου γεννήθηκα έχει ιστορία 12.000 ετών. Εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε τα της χώρας μας. Οι συνάδελφοί μας που εκπροσωπούν τους Κούρδους μίλησαν για την αυτοδιαχείριση στο, στο Χαλέπι. Έχουμε πόλεις με τοπικά συμβούλια. Έχουμε περιφέρειες, πολιορκία τώρα, που δεν λαμβάνουν ούτε προϊόντα, ούτε τρόφιμα, ούτε αλεύρι, τίποτα. Δεν είμαστε άγριοι. Η αγριότητα είναι χαρακτηριστικό του καθεστώτος. Έχουμε ανάγκη τα πάντα, αγαπητοί φίλοι. Χρειαζόμαστε τεχνογνωσία, γνώση. Ο λαός μας έχει ένα τεράστιο δυναμικό. Έχουμε ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν. Χρειαζόμαστε τεχνογνωσία, την τεχνογνωσία όλων των φίλων μας. Θα μιλήσουμε βέβαια τώρα και για την συνεργασία μεταξύ Εσμπολάχ και καθεστώτος. Έχω εδώ μια ερώτηση ο Μπασάρα Λασάντ θα εγκαταλείψει την εξουσία. Θέλει να διατηρήσει υπό την του ένα τμήμα του Συριακού εδάφους. Αληθεύει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το καθεστώς θέλει να ελέγχει ολόκληρη τη Συριακή επικράτεια. Αλλά έχει και ένα εναλλακτικό σχέδιο, δηλαδή να περιοριστεί στις ορεινές περιοχές και να εγκαταστήσει εκεί το καθεστώς του. Υπάρχει ένα θέμα πολύ σημαντικό. Μιλούμε για σύγκρουση μεταξύ Σουνιτών και Αλαουιτών και Σιητών. Εγώ γνωρίζω για επιστολές αλεβιτών στρατηγών που είναι αντίθετοι με το καθεστώς. φοβούνται ορισμένοι και το καθεστώς και τις άλλες θρησκευτικέ κοινότητες. Και το καθεστώς ζητεί από τους Αλεβίτες να τον υποστηρίξουν. Αν θέλει τώρα να εγκαταστήσει πολιτικό καθεστώς σε κάποιες ορεινές περιοχές, πρέπει πρώτα να προσελκύσει την υποστήριξη των Αλεβιτών. Αν αυτό βέβαια υλοποιηθεί, τότε ανοίγει η πηξίδα της Πανδώρας. Γιατί τότε να μην υπάρξουν χωριστά για τους Ρούσους, για τους Λιβανέζους και ούτω καθεξής. Ένα ξεχωριστό Εμμυράτο. Έχουμε και 2-3 εκατομμύρια Κούρδους στη Συρία. Έχουμε και Τουρκμένους. Τότε θα γίνει η Συρία θέατρο διαρκών συγκρούσεων που θα έχουν επιπτώσεις και για όλη τη διεθνή κοινότητα. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν είναι λογική. Ούτε έχει κανένα ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Υπάρχουν περιφέρειες των οποίων οι κάτοικοι θέλουν ένα μοντέλο αυτοδιαχείρισης. Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει με ειρηνικό τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να εξολοθρεύσουμε μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Το καθεστώς σκοτώνει του Σύρου γιατί δεν βρίσκει άλλη λύση. Οι Σύροι θέλουν απλώ να μπορούν να κοιμούνται χωρίς φόβο, να έχουν ελευθερία, ελευθερία έκφραση. Έχω ένα φίλο που ανήκε στον στρατό. Άκουσε ένα ανέκδοτο. Άκουσε ένα ανέκδοτο που διακομωδούσε τον πρόεδρο. Συμβαίνουν τα πράγματα αυτά. Και ποια ήταν η συνέπεια. Πέντε χρόνια φυλακή. Πέντε χρόνια φυλακή γιατί άκουσε το ανέκδοτο αυτό. Και δεν κάθισε αμέσως να γράψει έκθεση για να την υποβάλει στην Υπηρεσία Συλλογής Πληροφοριών της Αεροπορίας. Δεν υπάρχει χειρότερο καθεστώς από αυτό που ζούμε στη Συρία. Το καθεστώς νομίζω ψάχνει να βρει και εναλλακτικέ λύσεις. Για τους Κούρδους πριν από την εμφάνιση του κόμματος Μπαθ το 1963 η Συρία δεν γνώριζε ούτε εθνοτικά ούτε θρησκευτικά προβλήματα. Οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονταν πλέον για το ποιος ήταν Άραβας, Τουρκμένος, οτιδήποτε. Συμβιώναμε εν ειρήνη. Πήγαιναμε στο σχολείο χωρίς να ψάχνουμε να δούμε αν είμαστε μουσουλμάνοι ή χριστιανοί. Όποιος έχει επισκεφθεί την Συρία γνωρίζει καλά ότι ο Συριακός λαός ήταν λαός φιλόξενος που αγαπούσε τους άλλους. Ορισμένοι Αρμένοι μετά από τον πόλεμο ήταν, που ήταν ορφανά στη Δαμασκό οι οικογένειες υποδέχτηκαν τα ορφανά αυτά και τα έστελαν και στην εκκλησία. Μουσουλμανικές οικογένειες της Δαμασκού υιοθέτησαν ορφανά, μικρούς αρμενίους ορφανούς και τους έστειλαν στο σχολείο, Στην εκκλησία, συγγνώμη διότι θεώρησαν ότι είχαν χάσει την οικογένειά τους τα παιδιά αυτά και ότι οι Συριακές οικογένειες που τα υιοθέτησαν θα ήταν οι καινούργιες τους οικογένειες. Υπάρχει και η ιστορία του Αλγερινού Αμπτελκαντέρ που είχε υποδεχθεί 500 χριστιανικές οικογένειες. Δεν μιλούμε για αναγκαστική συμβίωση, αλλά για μια ειρηνική συμβίωση και ιδίω ως μουσουλμάνοι, ως μουσουλμάνος εγώ είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος όταν βλέπω ότι ο Ιησούς Χριστός έζησε εκεί, βάδισε στα χώματα αυτά. Υπάρχουν μονάχα δύο χωριά που μιλούν ακόμα τη γλώσσα του Χριστού. Δύο χωριά στη Συρία. Αυτό για μας είναι πηγή υπερηφάνειας. Το καθεστώς παρακινεί τους ανθρώπους να αλληλοσκοτώνονται. Και οι ηγέτες, θρησκευτικοί και μουσουλμάνοι και χριστιανοί, συμπαρατάσσονται με το καθεστώς. Και κάνουν το γύρο της Ευρώπης για να αποτρέπουν τον κόσμο να υποστηρίζει την αντιπολίτευση. Οι υπεύθυνοι ηγέτες των μουσουλμανικών και χριστιανικών θρησκευτικών κοινοτήτων. Οι ελεύθεροι υποστηρίζουν την αντιπολίτευση. Έχουμε προβλήματα με την κοινότητα των Λεβιτών που έχει γίνει όργανο του καθεστώτος. Εξ αντιθέτου, στη Συρία δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών. Βέβαια, ορισμένες, ορισμένα μέρη εκμεταλλεύονται τις διαφορές μας. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Τζον Κέρι και άλλους για να τους πω ότι δεν επιτρέπεται να γίνει πρόβλημα πραγματικό η διαφορά αυτή μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών. Και πριν λίγες μέρες ένας χριστιανός ιερέας δολοφονήθηκε. Εγώ βέβαια είμαι αντίθετος απόλυτα σε οποιαδήποτε δολοφονία. Εγώ θεωρώ ότι κάθε δολοφονία είναι βαρύτατο έγκλημα και υπάρχει τώρα κατακραυγή διεθνής μετά από την δολοφονία αυτή. Ένας μέγας επιστήμων ο μεγαλύτερος σύρος επιστήμων που δεν συμφωνώ με τις απόψεις του, ο δόκτωρ Σαΐντ Ραμαντάν, δολοφονήθηκε. Και το θέμα αυτό πέρασε στα διάφορα. Α, Κούρδος, κανένα θέμα να δολοφονηθεί. Αλλά έτσι και δολοφονηθεί ένας χριστιανός δίνεται υπερβολική έμφαση στο θέμα αυτό. Ενώ η ειρήνη πρέπει να ισχύει για όλο τον κόσμο και να φροντίσουμε να διατηρηθεί η ζωή όλων. Παλιά δεν είχαμε πρόβλημα. Το καθεστώς αυτό είναι η πηγή όλων των δεινών και των εντάσεων για μένα. για να βρεθεί πολιτική λύση ενδεχομένως χρειάζεται στρατιωτική επέμβαση. Για τη στρατιωτική επέμβαση όμως πρέπει να ληφθεί σαφής απόφαση. Να αποφασίσουν τα κράτη θα επέμβουν ή δεν θα επέμβουν. Διότι η κατάσταση επιτόπου αλλάζει καθημερινά. Σε λίγους μήνες και η στρατιωτική επέμβαση θα είναι μάλλον τελείως άχρηστη. Στην αρχή της αντίστασης Κανείς δεν ήταν ακραίος στη Συρία. Όταν ε, όμως ε, φάνηκε ότι η διεθνής κοινότητα επέτρεπε στο καθεστώς να κερδίζει χρόνο, ε, τότε περιπλέξαν τα πράγματα. Και, και τι θα πει στον κόσμο που βλέπει τα παιδιά του να σκοτώνονται, να τα σπάζουν, ε, ανθρώπους που έχουν δει τις μητέρες τους να βιάζονται. Υπάρχει ένας άνδρας που είδε το γιο του ε, να τον σφάζουν, να τον κατακρεουργούν, να τον ε, ακροτηριάζουν. Πού τον στέλνουν αυτόν, στην Αλκάιντα ή σε άλλα μέτωπα. Ε, έχουμε μια παροιμία εμείς που λέγει ότι, ότι ορισμένοι είναι αμήλικτοι και δεν αφήνουν ούτε στο Θεό τον ίδιο να, να πλαχνός απέναντι ε, σε άλλους ανθρώπους. Ποιος μιλάει σήμερα για το αίμα των παιδιών μας που χύνεται. Αυτό που μας απασχολεί είναι αν έχουν μούσει οι μουσουλμάνοι και όχι αν σφάζουν παιδιά θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και επιπτώσεις τους. Θα πρέπει όλη η διεθνής κοινότητα να στραφεί κατά του εξτρεμισμού. Βεβαίως, ε, αυτά είναι καταστροφικά φαινόμενα, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το κακό στη ρίζα του. Προσπαθώ να κινητοποιήσω τη διεθνή κοινότητα. Δεν θα πρέπει να υποστηρίζει η διεθνή κοινότητα δικτάτορες για τα συμφέροντά της. Πού είναι η ηθική της πολιτικής που ασκούμε. Χρειάζονται πολιτική με ήθος. Τα προβλήματα αυτά είναι αδιέξοδα και άλυτα. Ο συνάδελφος που θυμάται τη σφαγή στη Χάμα που είπε ότι ήταν τότε μαθητής ε, ήταν σφαγή 30.000 ε, και 40.000 και η διεθνή κοινότητα δεν επενεύει. Για ποιο λόγο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, οι πάντε ήταν ε, στο πλευρό του Χαφέζ Αλασάντ, του πατρός. Και τα συμφέροντα έχουν μεταβλητή γεωμετρία. Θα πρέπει πάντα να διαφυλάσσουν τα συμφέροντά τους εκατέρωθεν είτε υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον ε, ή ε, ε, είμαστε αντίθετοι στην κατάσταση. Όταν οι χώρες θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον τους να μην κάνουν τίποτα, γιατί θέλουν να διαφυλάξουν ορισμένες περιοχές για τα δικά τους ίδια συμφέροντα εις βάρος των συμφερόντων των λαών, αυτό θα έχει ολέθριες συνέπειες. Θέλω να αναφερθώ σε κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Γνωρίζω ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιες εντάσεις λόγω της παρουσίας ε, κάποιων κοινοτήτων, μουσουλμανικών κοινοτήτων. Γίνεται λόγος για την ταυτότητα. Και νομίζω ότι το βασικότερο πρόβλημα εδώ είναι ότι οι δικτατορικές κυβερνήσεις στον αραβικό κόσμο υποστηρίχθηκαν από την Ευρώπη και λόγω της καταστολής ε, στις αραβικές χώρες οι άνθρωποι έφυγαν από τις χώρες τους και ήρθαν να εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Και δεν έχουν ε, έτσι, ένα ευρύ πνεύμα αυτή. Ε, είναι ένα τμήμα της σκοταδιστικής κοινότητα στην Ευρώπη και είναι και πολιτικός οπορτουνισμός. Ορισμένοι θεώρησαν ότι μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη και ε, δεν θα έχει αυτό συνέπειες. Αλλά στη φυσική ξέρουμε ότι δεν πάει τίποτα χαμένο, καμία ενέργεια δεν χάνεται και στην πολιτική το ίδιο συμβαίνει. Δεν υπάρχει κενό. Όταν μιλάμε για ε, επίδραση των ε, ακραίων ομάδων, συχνά τίνουμε να υπερβάλλουμε τη σπουδαιότητά τους και τις συνέπειες. Θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να συνδέεται με το σεβασμό των ανθρώπων, με την αξιοπρέπεια. Η ταυτότητα μιας κοινωνίας έχει να κάνει κάνει με το δικαίωμα κάθε κοινότητας να αυτοπροσδιορίζεται. Βέβαια, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ας πούμε, στη Ρωσία έχει προτεραιότητα, διότι είναι ένα τμήμα της ρωσικής ταυτότητας. Υπάρχει ένα σύστημα στη Ρωσία που ε, φροντίζει να διαφυλάσει τους πάντες και καμιά φορά αναμειγνύονται διάφορα πράγματα. Θέλω να πω για τους Κούρδους ε, φίλους και αδελφούς μας από τότε που πήγα στο Πανεπιστήμιο έχω στενή ε, σχέση και επαφή με το κουρδικό ζήτημα. Αλλά υπάρχει και θέμα που έχει να κάνει με τις θέσεις των Κούρδων. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον κύριο Μασούτ Μπαρζανή και κάθε φορά που εμείς επιθυμούσαμε να αναγνωρίσουμε ε, κάποια οντότητα, παίρναμε αλληλογραφία από άλλες δυνάμεις και μας έλεγαν ότι εμείς είμαστε επίσημοι εκπρόσωποι των Κούρδων. Ο κύριος Μπαρζανή προσπάθησε να διοργανώσει στο Ερμπίλ πριν από ένα μήνα μια διάσκεψη για να βρεθεί μια λύση. Οι Κούρδοι πρέπει πρώτα απ' όλα να ενωθούν μεταξύ τους. Υπάρχουν προβλήματα και με το στρατιωτικό εμπάργο, τον εμπάργο όπλων στη Συρία και αλλού. Ορισμένες κουρδικές ομάδες υποστηρίζουν το κράτος σήμερα, ενώ κάποιε άλλες είναι αντίθετες. Ε, σε σχέση με αυτό εμεί και λόγω αυτού έχουμε δυσκολίε. Και το πρόβλημα είναι πρώτα πολιτικό και μετά εθνικό, εθνοτικό. Για τη συμμαχία ε, θα ήθελα να κάνω το εξή. τη δική μας. Είναι μια πολιτική οντότητα, δεν είναι κοινοβούλιο. Υπάρχουν χώρες άλλες που έχουν ασκήσει πίεση και ε, ε, υπήρξε άστοχη παρέμβαση έτσι ώστε η συμμαχία μας να γίνει κοινοβούλιο. Χωρίς εξουσία όμως, με ποια εξουσία. Εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των μελών της συμμαχίας μας αυτό μας ενδιαφέρει ή να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα. Χρειαζόμαστε βοήθεια, συμβουλές, πραγματογνωμοσύνη από τους φίλους μας. Ορισμένοι μπορεί να θεωρούν ότι είναι δυνατόν να λύνονται τα προβλήματα όλα των διαφόρων κοινοτήτων, των διαφόρων θρησκευτικών ομάδων, τον συνασπισμό μας, τη δική μας συμμαχία. Είναι πολιτική οντότητα, δεν είναι κοινοβούλιο αναγκαστικά αντιπροσωπευτικό όλων των δυνάμεων. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ε, ερωτήσεις σας. Ακούστε και κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ. Ότι στην Τύρο, Ταρτούς, οι περισσότεροι είναι αλεβίτες και ότι ορισμένοι που έφυγαν από τη Χόμς και από τη Χάμα πήγαν εκεί να εγκατασταθούν. Μα υπάρχουν και σουνητικά χωριά ανατολικά ε, της Χόμς που υποδέχονται αλεβίτες. Αλλά δεν ε, έχουν περικύκλωθεί χωριά χριστιανικά. Μην, μην πιστεύετε ότι διαβάζετε στο facebook. Δεν είναι όλα πληροφορίες διασταυρωμένες και επιβεβαιωμένες. Οι κουρδικές περιοχές έχουν αντιμετωπίσει μια κρίσιμη κατάσταση διότι έχουν φτάσει εκεί πολύ εκτοπισμένοι. Οι Κούρδοι είναι γενναιόδοροι από τη φύση τους και φιλόξενοι και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση όπως και κάτι και άλλων περιοχών. Καμιά περιοχή δεν γλιτώνει από αυτή την κατάσταση. Υφιστάμεθα τεράστιες πιέσεις. Ακριβώς λόγω της μετακίνησης των προσφύγων. Όποιος δεν συμφωνεί μαζί μας, όποιος θεωρεί ότι η Συριακή Επανάσταση ήταν σφάλμα, παρακαλώ να έρθει στη θέση των Σύρων. Για ελάτε στη θέση μας. Είσαστε σε μια δικτατορία, σε ένα καθεστώς εγκληματικό, σε μια εξουσία μαφία που ε, ε, καταστρέφει το σύνολο της χώρας. Το Στάλιγκρατ οχριά μπροστά στα όσα συμβαίνουν στη Σύρια και στην καταστροφή που ζούμε. Αν εσείς ζούσατε σε μια χώρα με τέτοια χαρακτηριστικά, τι θα κάνατε. Δείξτε μας το δρόμο αν ήταν σπάλμα η δική μας εξέγερση. Ευχαριστώ κύριε Μουάζελ Χατίμ. νομίζω πως όλοι εδώ έχουμε την αίσθηση ότι ακούσαμε, μάλλον μας δώσατε ένα πραγματικό χαστούκι για τους Ευρωπαίους που... Με την έννοια ότι μας υποχρεώνει η δική σας παρουσίαση να, μας, να δούμε την κατάσταση χωρίς προκαταλήψεις, επιφυλάξεις, να δούμε δηλαδή την βιαιότητα, ε, την ομότητα ε, αυτού του καθεστώτος, κατάματα. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Θα προσπαθήσουμε πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Ο κύριος Αλχατίμπη θα πρέπει νομίζω να γίνει δεκτός και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί κάποια θέματα ε, που συζητά το Συμβούλιο θα έπρεπε να ε, να συζητηθούν μετά από τη, ακούγοντας τη γνώμη του κ. Αλχατήπ και τη γνώση που έχει για τη χώρα και είχαμε την τιμή σήμερα να τον ακούσουμε. Έχουμε έναν ε, σπουδαίο πολιτικό ηθήνοντα που δεν ε, υπάρχει καμία αφιβολία, θα έχει και έχει και θα έχει και στη μετά Ασάντ εποχή ευθύνες μεγάλες, ηθικές και πολιτικές. Και έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Δεν βρήκαμε βέβαια λύση στο Συριακό. Αλλά είμαστε τουλάχιστον καλύτερα ενημερωμένοι και πιο έτοιμοι να ακούσουμε και να κάνουμε τις συζητήσεις με τα εκτελεστικά μας τις κυβερνήσεις, γιατί στην Ευρώπη σε αυτό το επίπεδο περιπλέκονται τα πράγματα, γιατί όπως σας είπα στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε ένα βαθμό Ε, συνένεσης που είναι στο ύψος ε, και που λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσει που εκφράσατε κι εσείς. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ να ζητήσω από τον Συμπρόεδρο αν θέλει κάτι να προσθέσει πριν κλείσουμε αυτή τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ κυρία Συμπρόεδρε. Ε, Όντως πιστεύω πως e, ve Türkiye parlamentosu burada ve Sayın Muaz El-Hatib'in söylediği Είμασταν παρόντε σήμερα εδώ όλοι και ο κύριος Αλχατίμπ είπε πολύ σημαντικά θέματα. Και Ελπίζω πως τα όσα υπόθηκαν δεν θα μείνουν μόνο εντός των ε, τυχών της αίθουσα, αλλά θα ακουστούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τον ευχαριστούμε για τον ηγετικό ρόλο που έπαιξε, που είπε τόσο ανοιχτά και ειλικρινά τα όσα γνωρίζει, την, μας δήλωσε τη θέση του. Ευχαριστώ την Ελένη. Και Κυρίως την ευχαριστώ που κάλεσε τον κύριο Αλχατίμπη σε αυτή τη συνεδρίαση. Χάρη σε ε, ηγέτες όπως εσείς είμαι, πεπισμένη, πως, είμαι πεπισμένος πως πολύ σύντομα τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν πρόγνωση για ένα εκατομμύριο πρόσφυγες ε, στην Τουρκία. Όχι, όχι, πρέπει να τελειώσει αυτή η υπόθεση πιο γρήγορα. Ένα ακόμα άτομο νεκρό σημαίνει θάνατο για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και θα πρέπει να ακουστεί η φωνή σας από σε ολόκληρο τον κόσμο ε, και όσο γίνεται πιο σύντομα ο κόσμος να γυρίσει σπίτια του να ζήσει με τις οικογένειες του, να γονείς με τα παιδιά τους μαζί. Κάναμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση χτες και σήμερα και ελπίζω Βέβαια, για κάποια δέντρα που κόπηκαν σε ένα πάρκο Είχαμε πολλούς πιο περισσότερους συμμετέχοντες ε, χτες, ε, ενώ εδώ που μιλάμε για χιλιάδες χιλιάδων νεκρούς ε, δεν συμμετείχαν τόσοι πολλοί. Πάντως ήταν ωφέλιμη συνεδρίαση και σας ευχαριστώ όλους. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και όλους, όλα τα μέλη της τουρκικής αντιπροσωπείας και όσους συμμετείχαν σε αυτή τη συνεδρία. ευχαριστώ.